Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, χρόνια πολλά, ιδιαίτερη χρονιά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θα διακόψουμε τις εργασίες μας πριν το τέλος του έτους. Θα είναι μια σύντομη χρονιά κοινοβουλευτική. Και μερικοί από εμάς θα ξεκινήσουμε την ε, προεκλογική μας εκστρέτεια. Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Πριέτο σε ό,τι αφορά την συζήτηση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πρώτα όμως να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Αλλά και πριν ακόμα τις ανακοινώσεις να σας ε, ενημερώσω για μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Θα γίνει μια αντιστροφή των σημείων 6 και 7. Δηλαδή, Πρώτα θα ενημερωθούμε για την πρόοδο των ε, τριμερών διαλόγων σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και μετά θα έχουμε την ανταλλαγή απόψε με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Απασχόλησης, της ΕΜΚΟ δηλαδή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις ε, μικρολέγες αυτές, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2 τώρα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Τρεις είναι οι πιο σημαντικές. Η πρώτη είναι μια επενθύμηση προς ε, τους ευρωβουλευτές και τους βοηθούς για να τους κινητοποιήσουν. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα που θα λάβει χώρα μεταξύ 20 και 22 Ιανουαρίου 2014. Δηλαδή θα διοργανωθούν δύο διακοινοβουλευτικές ε, διασκέψεις, τις οποίες θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικά Κοινοβούλιο. Το πρώτο αφορά το άρθρο 13 της ε, Συνθήκης Σταθερότητας ε, Συντονισμού και Διακυβέρνησης και η δεύτερη διάσκεψη αφορά το, την περίοδο 2013-2014, τον κύκλο δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το οριστικό σχέδιο προγράμματος θα μοιραστεί το συντομότερο δυνατόν. Πάντως η Επιτροπή Απασχόλησης ε, θα οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση στα πλαίσια αυτής της διακοινοβουλευτικής εβδομάδας την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και σας θέλω, παρακαλώ να έρθετε όσο περισσότεροι γίνεται, γιατί από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουμε πάνω από 140 βουλευτές. Έχουμε πολλούς εθνικούς βουλευτές, λοιπόν. Είναι σημαντικό να είναι αθρώα η προσέλευση και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, η έκτακτη συνεδρίαση που θα έχει διακοινοβουλευτικό χαρακτήρα στην Επιτροπή μας, η ΣΥΕΜ όπως λέμε στα αγγλικά, θα αφορά την ε, κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τα θέματα της απασχόλησης στα πλαίσια της ε, ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Σε συνεργασία με τους εθνικούς βουλευτές θα μιλήσουμε για τα θέματα της θέσπισης ε, της εγγύησης για τους νέους, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και το νέο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αυτόνομη έκθεση πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής μας με θέμα τα αποτελέσματα της Τρόικα, έκθεση δηλαδή Αλεχάνδρο Σέρκας, θα έχουμε την ευκαιρία για το θέμα αυτό και από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, που και αυτή θα συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας. Θα διοργανώσουμε λοιπόν μια κοινή ακρόαση, προκειμένου να ακούσουμε τους κοινωνικούς εταίρους την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, 3 με 4.30 το απόγευμα. Θα λάβετε ως ονούπο το πρόγραμμα αυτής της κοινή δημόσιας ακρόασης. Καταρχήν θα συμμετέχουν η Business Europe, η EDUC και η CIP που είναι ο φορέας ε, των επιχειρήσεων δημοσίων και κοινοφιλών υπηρεσιών. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν να έρθετε και σε αυτή την ακρόαση. Τρίτη σημαντική ανακοίνωση που αφορά το νομοθετικό μας πακέτο για την ε, έρευνα με δημοσκόπηση του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα και στην τελευταία μας συνεδρίαση, είχαμε καταλήξει σε συμβαστική λύση με τη Λιθωνική Προεδρία στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου της 17ης Ιανουαρίου και η συμβαστική αυτή λύση που αφορά κυρίως τις κατεξοδότησες πράξεις εξετάστηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων στις 20 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Δυστυχώς όμως η συμβαστική λύση που βρήκαμε με τη Λιθουανική Προεδρία απορρίφθηκε από την Κορεπέρ για τα κράτη-μέλη που ζήτησαν αναπομπή του φακέλου αυτού στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου για, τα, για τις στατιστικές. Του τέστην θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό με την Ελληνική Προεδρία. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να το φέρουμε στην Ολομέλεια για ψηφοφορία. περιμένουμε εξελίξει το Συμβούλιο, μία χειρονομία από το Συμβούλιο, γιατί στη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου τα σημεία που περιλήφθηκαν στη συμβαστική λύση για τις καταξιδότηση πράξης ήταν πολύ σημαντικά για μας. Και για να σας λίγο το υπόβαθρο και το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, Μα ενδιαφέρει ποιε είναι οι στατιστικέ που συγκεντρώνονται και το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν το περιεχόμενο αυτών των ε, στατιστικών πληροφοριών να προσδιορίζεται στι κατεξουδότητε πράξει, ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεμβαίνει στη διαδικασία. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό τμήμα του νομοθετικού μας έργου. Αυτά λοιπόν ως προς τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Σε ό,τι αφορά τη σε διερμηνία δεν ε, υπήρχε πρόβλημα. Κάθε φορά που ζητήθηκε η διερμηνία χρησιμοποιήθηκε και όλα. Επίσης υπάρχει αναμετάδοση από το web stream. Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου σας έχουν μοιραστεί. Και αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση, θα θεωρηθούν τα πρακτικά τη 10η Οκτωβρίου 25η-26 Σεπτεμβρίου 25 Σεπτεμβρίου 2013 ω εγκεκριμένα. Περνάμε τώρα στο σημείο 4, την εξέταση. Α, συγγνώμη, ο κύριο Σέρκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο ως προς τις ανακοινώσεις που μόλις τώρα κάνατε εσείς κυρία Πρόεδρε. Στη διακοινοβουλευτική εβδομάδα θα υπάρξει κάποια στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συζητήσει με τους συναδέλφους μας περί της έκθεσης για τις συνέπειες που έχουν τα προγράμματα της Τρόικας στις τέσσερις αυτές χώρες που έχουν εφαρμοστεί. Και εκεί δεν έχουμε συνδεθεί ε, Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το κοινωνικό σκέλος αυτών των προγραμμάτων σε αυτές τις τέσσερις χώρες. Αυτό ζητώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα μισάωρο μέσα στις ημέρες συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και οι συγητές θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τη σχετική έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Είστε σίγουρος, αγαπητέ συνάδελφα, Γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις εδώ. Είτε να γίνει στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής ε, συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΟΝ, είτε στην Ολομέλεια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον στα πλαίσια της Ολομέλειας που θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα. Οπότε θα φροντίσουμε εκεί να λάβετε το λόγο. Σε περίοπτη θέση μάλιστα. Στο επίκεντρο της διαδικασίας δεδομένη της ε, σημασίας που έχει το θέμα αυτό για την Επιτροπή Απασχόλησης. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Στο σημείο 4 θα εξετάσουμε τις 274 τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, για την έκθεση Σέρζιο Γκουτιέρες Πριέτο με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές τη ετήσιας επισκόπησης για, για την ανάπτυξη του 2014. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σέρζιο Γκουτιέρες Πριέτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, τις συναδέλφους της Επιτροπής μας. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, παρουσιάστηκαν 274 τροπολογίες. Άρα θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε συμβιβαστικές λύσεις και να εκπληρώσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει όταν αρχίσαμε να εξετάζουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μαζί με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Στόχος μας είναι λοιπόν να συντάξουμε μια έκθεση που να τύχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο. Στόχος μας είναι επίσης η έκθεση έκθεσή μας να μην είναι αντιφατική με την αντίστοιχη σχετική έκθεση της Επιτροπής ΕΚΟΝ και να υπογραμμίσουμε τα, τις επιδιώξεις οι οποίες πάντοτε χαρακτήριζαν ε, τη δική μας Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν περιθώριο ευέλικτο, ε, μεγάλο, για να πετύχουμε διαπραγματευτικέ λύσεις, συμβιβαστικέ. Θα πρέπει όμως να δούμε και το σημείο εκκίνησης. Πράγματι, ορισμένες πολιτικές ομάδες ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία και δίνουν διαφορετικές αποχρώσεις έννοιες ε, σε ορισμένα ζητήματα. αλλά και μέσα στο ε, κόλπους της ίδιας πολιτικής ομάδας υπάρχουν διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν και καλό όλους να επιδείξουν ένα πνεύμα συνεργασίας, να έχουν τη βούληση να πετύχουμε όλη συμβιβαστική λύση και να πετύχουμε και τους στόχους άλλωστε που μόλις τώρα σας παρουσίασα. Ένα παράδειγμα γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών, μπορούμε να πετύχουμε συμβιβαστικές λύσεις. Και λέω λοιπόν ότι συμφωνώ απολύτως με την κυρία Λόπεθ Φοντανέ, ε, με τις προθέσεις της υπέβαλε τροπολογίες για το ότι ας πούμε υπάρχει ανάγκη να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα πιο ευέλικτο ώστε να συγκεραστεί καλύτερα η δημοσιονομική εξυγίανση και προσαρμογή με την προστασία της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Άλλωστε αυτά είναι οι επιδιώξεις της δικής μας Επιτροπής. Συμφωνώ με την τροπολογία της ως προς τη βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Όμως, η διαφορά μας έγκυται κυρίως στους κοινωνικούς δείκτες. Ε, είναι ιστορική θέση της Επιτροπής μας, το πιστεύει και η κυρία Ντεμπάκερ, αυτή θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι κοινωνικοί δείκτες στο ευρωπαϊκό εξάμεινο να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους οικονομικούς δείκτες. Να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες των οικονομικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της οικονομικής διαδικασίας και πώς όλα αυτά πλήττουν την... και αυξάνουν τη φτώχεια, τον, κοινωνικό... τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην Επιτροπή μας δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε αυτές τις θέσεις και θα πρέπει να επιχειρηματολογούμε και να αγωνιζόμαστε ούτως ώστε οι κοινωνικοί δείκτες και όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν να είναι τουλάχιστον αντάξια ή να την χάνουν αντάξιας προσοχής με ε, τους οικονομικούς δείκτες και να συμφωνήσουν και να το συνειδητοποιήσουν και οι αρμόδιοι επί των οικονομικών στο Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα έχουμε την τροπολογία 176 η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη να μεταφέρονται ορισμένα δικαιώματα για τουλάχιστον τρεις μήνες σε σχέση με τους εργαζομένους που είναι αποσπασμένοι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχέση με το... είναι τροπολογία του Λαϊκού Κόμματος αυτού. Ωστόσο, στην προηγούμενη έκθεση της κυρίας Λόπεθ Φοντανέ σε σχέση με τα εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια την οποία θελήσαμε να, να υπογραμμίσουμε άλλωστε ήταν συμβαστική λύση της εισηγήτριας και τώρα θέλει να την καταργήσει και πρέπει να το σχολιάσω αυτό και δεν κατανοώ και τη θέση τη σε σχέση με όλες τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ε, τις ε, εκθέσεις σχετικά με την Πράσινη Βίβλο και τη Λευκή Βίβλο, την οποία, τις οποίες άλλωστε έχουμε στηρίξει στην ε, ε, Επιτροπή μας. Συμφωνώ με τις τροπολογίες της κυρίας Κορνέλησεν από την ομάδα των Πρασίνων, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τη δημοκρατική νομιμοποίηση. ό,τι έχει να κάνει με την ανάγκη επίτευξης διαθεσμικής συμφωνίας για να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όλο αυτό είναι απαραίτητο και πολύ καλώς το θέτει η κυρία Κορνέλισεν στην τροπολογία της. Την ευχαριστώ θερμά για αυτό. Έχουμε την τροπολογία 95 για τη σχέση μεταξύ φτώχειας και εκπαίδευσης. Συμφωνώ και πράγματι θα πρέπει να ενσωματωθεί αυτή η άποψη στην έκθεση. Αλλά και ε, την ε, προφύλαξη που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όταν μιλούμε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουν θετικές επιπτώσεις αλλά και παράπλευρες επιπτώσεις. και θα δουλέψουμε και πάνω στην τροπολογία 118 που ζητεί ίση μεταχείριση μεταξύ χωρών ή μεταξύ κυρώσεων των χωρών που έχουν έλλειμμα ημέν και πλεόνασμα ιδέ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι κυρώσεις να είναι αντίστοιχες και όχι μόνο να ε, πλήττουν τις ελληματικές χώρες αλλά και τις υπερβολικά πλεονασματικές. Ευχαριστώ θερμά τις ε, ε, προσπάθειες που κατέβαλε η ομάδα του Άλντε, την κυρία Χάρκιν, την κυρία Ντεμπάκερ κλπ. Πράγματι, με ενδιαφέρει ιδιαίτερο η άποψη του κυρίου Ντεμπάκερ μάλλον, με συγχωρείτε. Και νομίζω ότι συμφωνώ με τις τροπολογίες που έχει υποβάλει, οι οποίες προσθέτουν στοιχεία για την εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων, ε, για το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Με όλα αυτά μπορώ να συμφωνήσω. Κάτι το οποίο όμως ε, με εξέπληξε και νομίζω ότι εδώ διαφοροποιούμαστε ε, είναι οι τροπολογίες του που ζητούν να διαγραφούν πράγματα από την έκθεση. Θα ήθελα κύριε Ντεμπάκερ να μου εξηγήσετε ποια είναι η πρόθεσή σας, ποια, ποια είναι η πολιτική σκοπιμότητα να καταργηθούν οι συστάσεις που ζητάτε να καταργηθούν με την τροπολογία σας. Στην Επιτροπή ΕΚΟΝ δεν ε, συμπεριέλαβαν το παράρτημα των συστάσεων. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Από εκεί και πέρα. Έχουμε τα έτη 2008-2009, οπότε και ξεκίνησε η οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Και πράγματι έχουμε το σημείο κίνησης των κρατών μελών, κάτι το οποίο διευκόλυνε την έλευση της κρίσης. Είναι αληθές ότι δεν αξιοποιήσαμε την δεκαετία της ανάπτυξης από το 2000 και πέρα για να κάνουμε τις ε, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ε, και προσαρμογές στις εκάστοτε χώρες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μέχρι εκεί. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν οι συστάσεις αυτές. Θα πρέπει να ε, ε, ασκήσουμε κριτική π.χ. στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν είναι καθόλου ευέλικτο για την προσαρμογή του και την εξάλληψη του δημοσιονομικού ελλείμματος. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λοιπόν συνολική εικόνα για να είναι αντικειμενική η έκθεσή μας. Ευθύνη έχουν τα κράτη, σαφέστατα, αλλά αντίστοιχη ευθύνη έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει αυτό να το πούμε. Και να δούμε επίσης πώς θα εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις ε, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην αγορά εργασίας και κυρίως τις μισθολογικές αλλαγές. Είπαμε εξ αρχής ότι σαφέστατα πρέπει να μετριαστεί το εργασιακό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι Ορισμένες χώρες μπορούν πράγματι να γίνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές, ε, περικόπτοντας δραστικά το μισθολογικό κόστος, το μοναδιαίο. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Ε, βεβαίως συμφωνούμε όλοι αλλά όλες οι τροπολογίες που σκοπεύουν, αποσκοπούν στο να καταργηθεί αυτή η κριτική που ασκούμε στις χώρες οι οποίες περικόπτουν δραστικά το μισθολογικό κόστος, δεν είναι τροπολογίες που βοηθούν. Θα πρέπει να εξεταστεί αναχώρα η δυνατότητα αύξησης του ελάχιστου, ε, ε, του ελάχιστου ε, βασικού μισθού σε ορισμένες χώρες. Είναι κάτι που έγινε στη Γερμανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε. Αυξήθηκε κατά 10 δολάρια. Υπάρχουν χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, όπου ο βασικός μισθός είναι ο μισθός, ο μισός με συγχωρείτε, του βασικού μισθού που πρόσφατα θεσμοθέτησε η Γερμανία. Στην Ισπανία ας πούμε είναι 4 ευρώ την ώρα. Και είναι ζωτική σημασία σε αυτό για τις χώρες αυτές. Το να Το να καταργηθεί αυτή η τροπολογία χωρίς να δοθεί η δυνατότητα να μελετηθεί, να εξεταστεί, δεν είναι καλό σημείο κίνησης για να πετύχουμε συμβαστική λύση. Τέλος, θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι όλοι πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες και εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους μας ε, να είναι ισχυρή η έκθεση αυτή, να απηχεί το σύνολο της Επιτροπής μας και να συμπληρώνει την αντίστοιχη έκθεση των συναδέλφων μας από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στη Ρεζίνα Μπάστος που αντικαθιστά το σκιώδη συγγετή τη ε, Βερόνικα Λόπες Φοντανιέ, τη σκιώδη συγγετρία του ΕΛΚ. Ο, όταν α, ε, μας υπέβαλε ο εισηγητής στο σχέδιο εκθεσής του, ανέκυψε το ερώτημα το κατά πόσο είναι παραδεκτές κάποιες ε, παράγραφοι του αρχικού κειμένου. Και μάλιστα ε, ο εισηγητής συμφώνησε να τις τροποποιήσει κάπως για να γίνουν στο μεταξύ παραδεκτές. Και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι αυτές οι αρχικές παράγραφοι έδωσαν την ευκαιρία και σε άλλους συναδέλφους να πλειοδοτήσουν ή να συμβάλλουν στον προβληματισμό αυτό, προσθέτοντα κάποιους τομείς που εμφανώς ε, εκπίπτουν της αρμοδιότητας ε, της δικής μας Επιτροπής. Και εγώ επειδή είμαι αρμόδια για να βάλω μια τάξη στη δομή των εκθέσεων, θα πρέπει να κρίνω το παραδεκτό και κάποιων παραγράφων και κάποιων ε, τροπολογιών. Η Ρεζίνα Μπάστος που αποκαθιστά τη σκιώδη συγκέντρια του ΕΛΚ, την κυρία Λόπες Φοντανιέ. Ευχαριστώ. Όπως, ε, είπε και η, όπως είπατε η συνάδελφος Βερόνικα Λόπες Φοντανιέ, δεν ε, μπόρεσε να παραστεί, είχε ανελημμένες υποχρεώσεις στην εκλογική της περιφέρεια. Γι' αυτό και την αντικαθιστώ εγώ για... και θα παρουσιάσω τη θέση της για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σέρζιο Κουτιέρης Πρέτο για την έκθεσή του και θα σας διαβάσω το σημείωμα της κυρίας Λόπε Φοντανιά. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Είμαι βέβαιη ότι από την επόμενη εβδομάδα ήδη θα ξεκινήσουμε με επιτυχία τη διαπραγμάτευση για τις συμβαστικές λύσεις, γιατί ε, πολλές ε, από τις τροπολογίες έγιναν δεκτές από τον εισηγητή. Θα πρέπει πάντως, όπως και στο προηγούμενο εξάμεινο, να επιμείνουμε σε μια διαφοροποιημένη δημοσιονομική και φορολογική εξηγίαση που θα είναι αναλογική και θα προωθεί την ανάπτυξη. Οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς και είναι αυτή η στιγμή για να εξασφαλίσουμε την έξοδο από την κρίση και να επικεντρωθούμε στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι συντάξει είναι ένα από τα σημαντικά θέματα του κειμένου. Συμφωνώ με την τροπολογία 172 της ε, κυρίας ε, Ριόμεν Ρόιτεν που λέει ότι δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία δεδομένη τη συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σταξιοδοτικά δικαιώματα των επικουρικών συντάξεων καθώς και τις ε, δημογραφικές αλλαγές. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ενιαία, ένα ενιαίο όριο ηλικία ε, συντάξιμου και να περιοριστούν οι πρόορες δεξιοδοτήσεις. Άλλη, προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Επίσης θα πρέπει να επιτρέψουμε την εφαρμογή της αρχής ε, του front-loading και τη σωστή εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους. Για να προωθήσουμε λοιπόν την απασχόληση στους νέους θα πρέπει να μειώσουμε το φορολογική επιβάρηση της πρόσληψης των νέων ή να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους δίνοντας φορολογικά ενάψματα. Επίσης θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την εκπαίδευση με τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Επίσης με την ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι άλλο νευραλγικό σημείο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίξαμε και το πρόγραμμα COSME και τον ορίζοντα 2020. Θα θέλαμε όμως να τεθεί ένα τέρμα στον κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τέλος, η συνάδελφος Λόπε Φοντανιέ ε, τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να μειωθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σας ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ, Μαρία Άλισον και στη συνέχεια Ντεμπακέρ. Υπεύθυνος για την ε, ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής Επιτροπής. Κυρία Άλισον, ευχαριστώ πολύ. Uh, κυρία Κορνέλισεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγήτρια, τους, τις εισηγήτριες. Ξέρω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την ασυμβατότητα μεταξύ των δύο εκθέσεων και να έχουμε μια ευτυχή έκβαση χαίρομαι ε, που υπάρχουν και οι δύο πλευρές γιατί δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμες ε, οι απόψεις μεταξύ των εισηγητών. Ε, πιστεύω όμως ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ παραγωγικά μεταξύ μας. Υπάρχει το έβριμα ε, της δημοκρατίας και του πώς ε, θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και τα κοινοβούλια. Όλοι ζητούμε μεγαλύτερη ανάμειξη του δικού μας κοινοβουλίου, για παράδειγμα, ε, και στην ετήσια έρευνα για την οικονομία, αλλά καμιά από τις προτάσεις μας δεν έτυχε ευνοϊκής αποδοχής και νομίζω ότι πρέπει να υποβάλουμε ένα ισχυρό και συγκεκριμένο για μια διοργανική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Αυτό ε, θα είναι ένας τρόπος ενίσχυσης ε, της δημοκρατίας χωρίς πραγματική αλλαγή των συνθήκων και χαίρομαι που οι συγητές συμφωνούν μαζί μου. Επίσης συμφωνώ ότι οι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι και να διασυνδέονται με τους οικονομικούς δείκτες δεν θα βοηθήσει και πολύ αν παραμείνουν ε, ανεξάρτητοι, χωριστοί. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να γίνουν περικοπές στο κόστος της περίθαλψης, ε, το κόστος πρέπει να περικοπεί κατά τρόπο που να μην πληγεί η καθολική κάλυψη του πληθυσμού, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνικοί δείκτες να, διαμορ... να συνδιαμορφωθούν και από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια τρομπολογία, η 82, την οποία υποβάλαμε κατά την ε, Υπουργική Συνάντηση. οι Υπουργοί θα συναντηθούν και προτείνει ε, ο εισηγητής να το εξετάσουν. Νομίζω όμως ότι οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Υπουργοί για την Κοινωνική Πολιτική πρέπει να συναντηθούν από κοινού, γιατί οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να είναι παντού παρούσες. Δεν είναι δυνατόν οι κοινωνικές και οι οικονομικές πολιτικές να είναι χωριστές. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να, να υπάρξει κοινή συνάντηση μεταξύ των ε, δύο πριν από την τελική συνάντηση. Επίσης, ε, θα ήθελα να ψηφίσουν όλοι υπέρ της 118 τροπολογίας. Πρόκειται για την, το τρόπο αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανα, ανισορροπιών. νομίζω ότι πρέπει να, είναι, να υπάρχει μια προσπάθεια για συμμετρικότητα και δικαιοσύνη γιατί διαφορετικά πλήττεται γενικά η ισορροπία και το έλλειμμα. Υπάρχει, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί αυτή η ιδέα της συμμετρίας και της δικαιοσύνης. Και τελικό σχόλιο, σχετικά με την τροπολογία 154. Ε, ζητούμε και πάλι από τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν ε, σχέδια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, συνοδευτικά προς τις εθνικές τους μεταρρυθμίσεις. Πριν από αρκετά χρόνια είχε ξαναζητηθεί αυτό και κανένα κράτος μέλος δεν υπέβαλε τέτοια σχέδια. Είναι καταθλιπτικό που πρέπει να το ζητούμε ξανά από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι η ανεργία των νέων και η ανεργία γενικότερα δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με μέτρα ενεργοποίησης και κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή και προοδευτική έκθεση. Ξέρω ότι έρχονται οι εκλογές, αλλά νομίζω ότι ειδικά για αυτήν την έκθεση επειδή πρέπει πραγματικά να στείλουμε ένα ισχυρό σήμα ως κοινοβούλιο συνολικά, ας παραμερίσουμε λιγάκι τις ε, ιδέες του καθενός και ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ευρύτερη πλειοψηφία. Πρόεδρος, ευχαριστώ για αυτήν ε, την ε, αξιολόγηση, για αυτά που μέλη να γίνουν στο Κοινοβούλιο, ε, την παραμονή των ευρωεκλογών. Φιλ, εκ μέρους της ε, Οικονομικής Νομισματικής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ε, καλή χρονιά. Πιστεύω θα είναι μια συναρπαστική χρονιά. Καλή τύχη σε όλους. Ε, βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ καλή παρουσίαση της έκθεσης με την έκθεση παρουσίασης που έγινε. προχωρούμε τώρα στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια των προηγούμενων ομιλητών. Πραγματικά πρέπει να να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Στο παρελθόν πιστεύω ότι υπήρξαν πολλές αντιφάσεις και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ζητώ συγγνώμη που ο συνάδελφος δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Ε, να προσπαθήσω να απαντήσω και σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μου απέθυναν οι συνάδελφοι και να πω κάτι και για τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Οφείλω να πω ότι στην Επιτροπή μας ε, το, η δουλειά έχει προχωρήσει αρκετά. Ε, υπάρχει ευρεία συνένεση για τα περισσότερα από τα θέματα που θίγονται στην έκθεση αυτή. Ε, και αυτό προσπαθώ να το λαμβάνω υπόψη μου όταν ε, στο επόμενο ραντεβού μας και με την Επιτροπή Απασχόλησης να δω να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα μεταξύ των δύο εκθέσεων. Φυσικά υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές απόψεων, υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο που βλέπει ο καθένας την κρίση και διαφορές και ως προς τις λύσεις. Και αυτό πιστεύω ε, αντανακλάται στη θέση των εισηγητών και στις θέσεις των τροπολογιών της δικής μου ομάδας και των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Για μένα η κρίση αυτή, η οποία συνεχίζεται για πέντε συναπτά έτη πλέον, μπορεί να επιληθεί μόνο εάν έχουμε μια, ένα πολύ σαφές όραμα και διακρίνουμε ξεκάθαρα το δρόμο που πρέπει να πάρουμε. Νομίζω ότι μεγάλο φταίξιμο έχει και η Επιτροπή. Η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο έχει συντάξει ένα πλαίσιο για την οικονομική σταθερότητα. Ε, η ομάδα μου το στηρίζει αυτό, θεωρείται το πλαίσιο αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα και μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ελαφρύνουν τις πιέσεις που υφίστανται και εξασφαλίζει ότι η μη επανάληψη κάποιων από τα σφάλματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε αυτή την ελαφρά ανάκαμψη, πολύ εύθραυστη, πολύ πρόημη στην Ευρωζώνη. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι, συμφωνώ. Από την άλλη να μην είμαστε και υπερβολικά απεσιόδοξοι. Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Όταν μιλούμε για προσαρμογές, μιλούμε φυσικά για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αυτό αντανακλάται και σε αυτήν την έκθεση. Υπάρχει η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών αγορών, των, συνταξιοδο... των συστημάτων συνταξιοδότησης, της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών. Όλα αυτά τα μέτρα βέβαια πρέπει ή θα έπρεπε να εστιάζονται στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να, να σημειωθεί πρόοδος. Ε, για μας αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να δούμε ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα, θέλουμε να δούμε ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος μακροπρόθεσμα για να ε, έχουμε επαρκή ανάπτυξη, επαρκή μεγένθεση, επαρκή θέσεις εργασίας στην Ευρώπη για τους λαούς. Και βέβαια η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που διαθέτουμε για να υπάρξει αυτή η οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Υπάρχει και όλη η συζήτηση για τη μείωση του χρέους. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή και στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Πολλά μένει να γίνουν ακόμη. Έχουμε τους ε, τραπεζικούς ισολογισμούς. Πολλά μένει να γίνουν εκεί. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία για να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι θα έχουμε τις προοπτικές αυτής της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, χρειάζονται λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις και πρέπει να τις στηρίξουμε. Όταν μιλούμε για το χρέος και την ανάπτυξη, όλοι γνωρίζουμε ότι πολλή ανάπτυξη προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαίρομαι που η έκθεση το τονίζει αυτό, που υπάρχει ειδική μνήα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ ήμουν συντάκτης μιας πρωτοβουλία, ίδιας πρωτοβουλίας ε, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χαίρομαι που πολλά από τα εργαλεία που παρέχει η Κομισιόν υλοποιούνται στα κράτη-μέλη τώρα. Χαίρομαι πολύ. Ε, βεβαίως, ε, μιλούμε πάντοτε και για την ε, απασχόληση, την ανεργία, την ανεργία των νέων. Πραγματικά πρέπει να εστιάσει η συζήτηση και σε αυτό, όπως το κάνει η έκθεση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη και καλύτερη εκπαίδευση, ε, πρωτοβουλίες στην αγορά εργασίας που θα διασφαλίζουν ότι οι άνεργοι θα επιστρέφουν στην απασχόληση όσο το δυνατόν δυνατότερα. Σε πάρα πολλές χώρες υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις της εργασίας η μεταρρύθμιση εργασίας πιστεύω πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη πέρα από τις διαφορές απόψεων που έχουμε. Πρέπει να είναι πιο εύκολο για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να βρίσκουν τόπο συνάντησης, αλλά και πρέπει να εξατομικεύεται η κατάσταση στις επιθυμίες και στις ανάγκες των ανθρώπων. Τα συστήματα που βλέπουμε σήμερα σε πολλά κράτη-μέλη ε, δεν επιτρέπουν τις αναγκαίες προσαρμογές. Όταν μιλούμε για την ανεργία των νέων, αυτό συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για τη φτώχεια. Ε, ο πιο σημαντικός τρόπος να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια είναι να επανέλθει ο κόσμος στην αγορά εργασίας. Αυτό νομίζω είναι χρειάζεται αυτή η ενεργηγός συμμετοχή στην εργασία. Αυτό είναι που συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Και έτσι έρχομαι και στη συζήτηση για τους Κοινωνικού δείκτες. Και επανέρχομαι στο πρώτο μου σχόλιο. Είχαμε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και τώρα θέλουμε να σταθεροποιήσουμε και τα κοινωνικά συστήματα σε πολλά κράτη-μέλη. Είχαμε τόσα πακέτα. Πρέπει να δώσουμε σε αυτό το πλαίσιο τη δυνατότητα να υλοποιηθεί με σαφείς στόχους, με σαφείς φιλοδοξίες, με συγκεκριμένα κριτήρια. Ε, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συζήτησης, αν θέλετε. Εδώ η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στην πιο συγκεκριμένη υλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά σχόλια. Υπάρχει και η συζήτηση για την δημοκρατική νομιμοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ στην Επιτροπή μας πρέπει να υιοθετήσουμε μια ισχυρή πολιτική θέση. Τα εργαλεία που έχουν τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα για να ξαναμπούμε στο δρόμο προς την ανάπτυξη ε, για αυτό για να γίνουν αυτά, η ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας είναι πραγματικά ουσιώδης και ελπίζω με τους συναδέλφους και με τους πρασίνους και με άλλους να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να εξασφαλίσουμε ως κοινοβούλιο ότι θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Δύο λόγια για το παράρτημα. Πολύ θερμή συζήτηση ε, ε, έγινε τις τελευταίες δύο συζητήσεις είναι πολύ σαφές σε μένα. Συμμετείχα και στο παρελθόν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε εκτεταμένη συνένεση για αυτά τα ε, για το παράρτημα που περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις προς την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Και γιατί είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η δυσκολία, γιατί υπάρχουν οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων. Οι συστάσεις αυτές απαιτούν μεγάλη, πολύ μελέτη, πολύ προσοχή, χρήση το, της σωστής διατύπωσης, να, είναι, να δώσουμε τις σωστές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, προς το κάθε κράτος μέλος. Είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς ε, γενικού περιεχομένου δηλώσεις από ότι συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στην ε, ΕΚΟ και αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε με τα παραρτήματα, να έχουμε πολύ συγκεκριμένες εκθέσεις με ισχυρή, με ισχυρή διατύπωση και να στείλουμε ένα πολύ σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα με την ίδια την έκθεση. Νομίζω ε, ως προς τις συστάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ομοφωνία. Για τα πλεονάσματα, για παράδειγμα. Ε, μια χώρα που έχει πλεόνασμα, που είναι εύρωστη οικονομικά, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν τις συνέπειες τους, αλλά οι χώρες που τα πάνε καλά να μπουν στο, στην ίδια βάρκα μαζί με τις άλλες που δεν τα πάνε καλά, νομίζω δεν είναι και τόσο λογικό αυτό. Μάλλον λοιπόν δεν θα προχωρήσει το ζήτημα με τα παραρτήματα. Θα το συζητήσω και με τους σκιώδεις εισηγητές. Γι' αυτό και έχω υποβάλει και μια τροπολογία να μην συζητήσουμε τα παραρτήματα αυτή τη στιγμή, Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό να έχουμε μία συγκεκριμένη, ξεκάθαρη ε, έκθεση με τη σωστή ισορροπία μεταξύ του κοινωνικού και του οικονομικού τομέα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τα συγκεκριμένα παραρτήματα. Έχω υποβάλει ήδη κάποια σχόλια προς τους συζητητές. Ελπίζω και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ε, μείναμε λίγο πίσω στην ώρα, αλλά μια και είναι τόσο σημαντική η συζήτηση, θα ήθελα να κάνω δύο διαδικαστικές παρατηρήσεις και μία παρατήρηση επί της ουσίας, ό,τι αφορά τα διαδικαστικά. Ο κύριος Ντεμπάκερ μας είπε ότι τα παράρτηματα αφορούν κάποιες λεπτομέρειες που θα καταστήσουν πιο δυσνόητο το κείμενο ή θα εμποδίσουν την επίτευξη συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνω ότι κάποιες πολιτικές ομάδες, ιδιαίτερα η δική μου, ε, έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα της ετήσιας επισκόπηση για την ανάπτυξη. Και μάλιστα ζήτησαν και από φορείς πέραν της σφαίρας των Βρυξελών να κάνουν κάποιες αναλλακτικές τέτοιες αιτήσει επισκοπήσεις για την ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να αναθέσει την εκπόνηση τέτοιων μελετών σε, άλλους φορείς. Γιατί πάσχουμε από δημοκρατικό έλλειμμα. Και από την αρχή είδαμε ότι η οικονομική πολιτική της Ένωσης γίνεται με βάση την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δίκιο έχετε κύριε Ντεμπάκερ, ότι όλα αυτά στηρίζονται σε μελέτες, σε πυρογνωμοσύνη σημαντική και ότι χρειάζονται κάποια στοιχεία από άλλους φορείς, από άλλους εμπειρογνώμονες. Αυτό έκαναν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, η δική μου πολιτική ομάδα και θα ήθελα να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπησέλθει στο σκληρό πυρήνα των συστάσεων Όλη η προεργασία που έγινε και όταν λέω από εμά εννοώ από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Ανάπτυξης και από την Επιτροπή Απασχόλησης και πριν ακόμη τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είτε για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, είτε για τους βασικούς προσανατολισμούς για την οικονομική πολιτική. Όλες αυτές οι προσπάθειες έγιναν υπό την ευθύνη του Τζάμπα Όρη όταν συζητήσαμε τι κατευθυντήριε γραμμέ για την απασχόληση. Αν δεν λάβουμε όλα αυτά τα πράγματα σοβαρά υπόψη, τότε δεν θα έχουμε λόγο σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προσδιορισμό του πλαισίου και του συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Ενώ σε μια δημοκρατική κατάσταση είναι η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο εργαλείο για τον προσδιορισμό του κοινωνικού συμβολέου. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και προτείναμε να περιλάβουμε στο παράρτημα τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις τροποποιήσουμε και ελπίζω να δημιουργηθεί ε, η κρατούσα γνώμη στην Επιτροπή μας και μια πλειοψηφία για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερη διαδικαστική παρατήρηση. Εδώ θα ήθελα να ομολογήσω την αδοημοσύνη μου, γιατί πολύ ακροθυγός ε, κοίταξα αυτές τις 274 τροπολογίες που υποβλήθηκαν για την έκθεση του Σέρζιο Γκουτιέρες Πριέτο ε, και προβληματίστηκα κυρίως από ένα θέμα. Τη στιγμή ακριβώς που θα ξεκινήσουμε την προεκλογική μας εκστρατεία, ε, φαίνεται ότι η συνέχεια των εργασιών που ξεκίνησε ο Βανερόν Πόη θα συνεχιστεί θα προχωρήσει και θα, ίσως υπάρξουν και νέες εξελίξεις. Και πέραν του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσαμε να έχουμε εργασίες και με πρωτοβουλία του Συμβουλίου για την εμβάθυνση της ΩΝΕ και μάλιστα σε μια περίοδο που το Κοινοβούλιο θα είναι αδρανές. Οπότε καλό θα ήταν επ' ευκαιρία τη εξέταση τη αιτήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου στην Ολομέλεια να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή η κοινοτική μέθοδο ε, στην προσπάθεια εμβάθυνση τη ΟΝΕ. Και οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Συμβουλίου κατά την περίοδο που το Κοινοβούλιο θα είναι κλειστό θα πρέπει να επανεισαχθεί και μετά τις εκλογές ε, και να εξεταστεί στα πλαίσια της κοινοτικής μεθόδου. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Στα κράτη-μέλη στυλιτεύουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και προσπαθούμε να το γεφυρώσουμε ταυτόχρονα παραγωνίζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι το α και το ω των πάντων, αλλά σε πλαίσια, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δημοκρατικής νομοποίησης νομίζω ότι είναι το καλύτερο φόρουμ για την πραγμάτωσή της. Τώρα για τα πλεονάσματα που έχουν ορισμένε. χώρες. Σίγουρα δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους ενάρετους. Αλλά οι ενάρετοι και οι αρετοί δεν νοούνται μεμονωμένα και υπάρχουν χώρες που έχουν πλεονάσματα Φυσικά γιατί τα αξίζουν και γιατί έχουν πολλές αρετές και πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσονται αυτές οι χώρες σε ένα πλαίσιο που εμ, εποφελούνται από αυτή τη γενική ενισορροπία. Οπότε δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη το πλεόνασμα ορισμένων χωρί να λαμβάνουμε υπόψη και τη γενική ενισορροπία. Σίγουρα και οι χώρε που έχουν έλλειμμα θα πρέπει να κάνουν προσπάθειε, αλλά δεν μπορούν από μόνε του να λύσουν το πρόβλημά του. Γιατί δεν είναι μεμονωμένο αυτό το έλλειμμα. Το έλλειμμα μερικών δημιουργεί το πλεόνασμα άλλων. Και αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Και λυπούμε πραγματικά που έχει περάσει τόσο καιρό, αλλά ε, δεν έχουμε ακόμη καταλήξει μια συμφωνία. Κύριε Σιγητά, θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσετε στα σχόλια των συναδέλφων και να σας θέλω παρακαλέσω να είστε πιο σύντομος ε, αυτή τη φορά. Και είμαι βέβαια ότι θα τα καταφέρετε. Βεβαίως κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, όπως μου υποδείξατε. Να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Κορνέλισεν, την κυρία Μπρές, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τη Δημοκρατική Νομιμοποίηση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το πώς εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τι έχει συμβεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια που ε, έχουμε θεσμοθετήσει αυτή τη διαδικασία. Είχαμε άμεση μεταφορά κυριαρχίας εθνικής σε θεσμικά ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν αυτό δεν συνοδευτεί με μεγαλύτερο, από μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο κυρίως από αυτό το κοινοβούλιο, τότε αυτή η διαδικασία θα χωλαίνει και τελικά θα νομίζουμε ότι εξυπηρετούμε τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά ουσιαστικά θα υπονομεύουμε τις δημοκρατικές εγγυήσει που του παρέχουμε και που ε, ε, ενσαρκώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εθνικά μετερρυθμιστικά σχέδια με την έγκριση του εξάπτυχου πέρσι του Sixpack είναι δεσμευτικά. Σαφέστατα. Άρα ή θα ενισχύσουμε την άποψη, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία ή όταν ή αν κάποια κράτη-μέλη δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοκρατικής νομιμοποίησης, ε, το, υπάρχει πρόβλημα διότι δεν θα έχουν συνομιλήσει με όλους τους κοινωνικούς φορείς και γι' αυτό ε, χωλαίνει και ιστερεί από πλευρά δημοκρατικής νομιμοποίησης αυτή η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει λοιπόν η έκθεσή μας να είναι συμβατή με την έκθεση της ΕΚΟΝ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αντιγραφή της, να τη μιμούμαστε σε καμία περίπτωση. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα εξετάσει το θέμα από τη δική της σκοπιά. Και σαφέστατα οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι πολύ καλύτεροι από τους, από τους κοινωνικούς δείκτες και τους δείκτες απασχόλησης. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε τόσο θετικοί όσο η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η απασχόληση ε, μειώνεται. Η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης μειώνεται επίσης των προσφερόμενων, των όποιων. Και άλλωστε σε πολλές χώρες ε, τρεις στους τέσσερις νέους βρίσκονται εκτός απασχόλησης για άλλη μια ε, χρόνια. Υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει φτώχεια μεσοπρόθεσμη, όλα αυτά είναι σαφέστατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε νοικοκυριά τα οποία ε, κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού και ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά είναι στοιχεία τρομακτικά και δείχνουν ότι δεν πρέπει ως Επιτροπή μόνο να εκφράζουμε αισιοδοξία. Δύο είναι οι πραγματικότητα. Είναι μια η πραγματικότητα της βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου, ε, της εξάλληψης σταδιακά του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Όλα αυτά τα θετικά υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και δεν μπορούμε να, να κλείνουμε τα μάτια σε αυτήν. Λοιπόν, ε, η έκθεσή μας πρέπει να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα. Επιμένω λοιπόν το να έχουμε μια ε, έκθεση συμβατή με αυτή της ΕΚΟΝ δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια έκθεση που να είναι αντιγραφή ε, της έκθεσης της ΕΚΟΝ. Δεν θα πρέπει να τιμιμούμαστε. Και δεν λέω ότι η Επιτροπή φταίει για όλα κύριε Ντεμπάκερ. Σίγουρα υπήρξε μεταφορά εθνικής ε, κυριαρχίας για διάφορα οικονομικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο όρισαν το χρονοδιάγραμμα προσαρμογής και εξάλληψης του εθνικού ελλείμματος του εκάστοτε. Ορισμένες μελέτε μελέτες υποστηρίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό έπληξε πολύ περισσότερο την απασχόληση επειδή ήταν τόσο στενό παρά τα καλά που έφερε. Και αυτή η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που έπρεπε να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στραγγάλισε την απασχόληση, στραγγάλισε τις οικονομίες ε, στις ε, χώρες μέλη και δεν επέτρεψε στις χώρες μέλη να βγουν από την κρίση. Αυτό είχε ε, πολύ μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο από την εργασιακή μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα ή δεν έλαβε χώρα σε ορισμένε χώρε μέλη. Σαφέστατα ε, είναι ανάγκη να κάνουμε κοινωνικέ μεταρρυθμίσει και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Με ποιο κοινωνικό κόστο όμω, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς Σαφέστατα, ε, ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζονται ε, με συγκεκριμένο τρόπο και ορμώνται από συγκεκριμένο εφαλτήριο, αν θέλετε. Και όλοι το βλέπουμε αυτό. Έχουμε πολύ ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Όλα αυτά υπάρχουν στα παραρτήματα και τελικά σε κάθε σύσταση αναχώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που έκανε ήταν αντιγραφή και επικόλυση ε, της ίδιας διατύπωσης, της ίδιας παραγράφου. Λες και είναι το ίδιο ε, το εκάστοτε π.χ. συνταξιδοτικό σύστημα της Ισπανίας με το αντίστοιχο της Ουγγαρίας, για παράδειγμα. Μην είμαστε αφελείς πολιτικά, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανακτήσει πλήρως το ρόλο που του αναλογεί, να τον διαδραματίσει πλήρως. Είναι κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή που οικοδομούμε την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει τη θέση του ως πολύ σημαντικού παίκτη γιατί είναι άλλωστε και το μόνο όργανο που χαίρει της δημοκρατικής νομιμοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στις 22 Ιανουαρίου και θα τις ψηφίσουμε την επομένη, δηλαδή στις 23 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή ταυτόχρονα με την έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ ε, για την Επιτροπή ΙΑΕΚΟΝ στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Καλώς. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας μας διάταξης. Και καλούμαστε λοιπόν να ε, ξεκινήσουμε τη δημόσια ακρόαση σχετικά με τις πτυχές απασχόλησης και κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των δράσεων της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης που υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Αλεχάνδρο Θέρκας και έχουμε τέσσερις διακεκριμένους προσκεκλημένους. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι ε, ξεκινούμε τις εργασίες με λίγη καθυστέρηση. Εσείς οι τέσσερις ε, προσκεκλημένοι μας ε, παρακολουθείτε τις εργασίες μας από την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας και έτσι έχετε μπει πλήρω στο πνεύμα ε, του διαλόγου που κάνουμε εδώ. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Χωσέ Σίλβα Πενέδρα, κύριε Ρέιμον Τόρες, κύριε Πέτρο Στάγκο και κύριε Θόρστεν Σούλτεν, θα ήθελα καταρχάς εν συντομία να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Θέρκας για να μας πει δύο λόγια για το πνεύμα που τον διείπε κατά τη διάρκεια των εργασιών του, αλλά και για να σας θέσει ενδεχομένως ορισμένα, ορισμένες ερωτήσεις κέρυες, οι οποίες αφορούν, έχουν σχέση με τη δική μας δημόσια ακρόαση. Μία ακρόαση που εντάσσεται σε ένα πιο ευρύ ε, πλαίσιο. Έχουμε ακρόαση λοιπόν επιρογνωμόνων, ειδικών σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως σας είπα και προηγουμένως, να έχουμε ε, κοινή εξέταση με τα μέλη της ε, Επιτροπής Οικονομικής και, Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων για να εξετάσουμε όλα τα θέματα. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά το ανώτερο. Ευχαριστώ να καλωσορίσω πρώτα θερμά τους εμπειρογνώμονές μας και να τους ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία τους εδώ ε, και θα μας βοηθήσουν στο έργο μας που θα είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου γιατί οι ιστορικές εξέλιξεις μας ε, φέρνουν να δίνουμε εξετάσεις μπροστά στους Ευρωπαίους πολίτες και θα πρέπει όλα τα κοινωτικά θεσμικά όργανα να δώσουν λόγο να γίνουν υπόλογοι και να δώσουν και εξηγήσει για τι δραστηριότητε του. Διανύουμε την σοβαρότερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουμε τεράστιους κλονισμούς και κλειδονισμούς και σημαντικά προβλήματα όχι μόνο για τους ιδιώτες αλλά και για το ολόκληρο το σύστημα και διανύουμε μια ιστορική στιγμή και θα πρέπει με θάρρος και χωρίς φόβο να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Γιατί δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να περιγράφουμε μια ιδηλιακή κατάσταση, να έχουμε μια σοβαρή και ανησυχητική κατάσταση και φοβερά ρήγματα και στην Ευρώπη και στους Ευρωπαίους πολίτες και σοβαρούς τριγμούς. Όπως είπε η, ε, πρόεδρός μας, ε, η έκθεση αυτή θα έχει και μια οικονομική πτυχή ε, και αυτή θα την αναλύσει η Οικονομική Επιτροπή, αλλά και κοινωνικές πτυχές και πτυχές απασχόλησης ε, και αυτές θα τις αναλύσουμε εμείς. Βρισκόμαστε στη φάση της εξέτασης των ε, τροπολογιών και στο διάλογο που έχουμε με την κοινωνία των πολιτών. Γιατί θέλουμε μια δημοκρατική συζήτηση και μια ανάλυση για να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι κοιτάζουμε κατάματα την πραγματικότητα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να ξεπεράσουμε αυτά τα τρία τραγικά χρόνια που μόλις περάσαμε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα δύο κεντρικά σημεία της έκθεσης. Καταρχήν, ε, εμείς περιοριστήκαμε στις κοινωνικές πτυχές, γιατί η Οικονομική Επιτροπή θα ασχοληθεί με τις πιο διαρθρωτικές διαρθρωτικές πτυχές των προγραμμάτων της Τρόικα και επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις χώρες, σε αυτές που υποβλήθηκαν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν εξετάζουμε την κατάσταση στην Ισπανία ή άλλων προγραμμάτων χωρών βοήθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά περιοριζόμαστε μόνο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Στις χώρες δηλαδή που εφάρμοσαν προγράμματα διάσωσης δημοσιονομικής προσαρμογής. Εδώ έχουμε και επιθυμούμε δύο πράγματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο απολογισμός από πολλά κοινωτικά θεσμικά όργανα. Βγήκε η Ιρλανδία, βγήκε η Ισπανία από το σύστημα, φαίνεται ότι θα βγει και η Ισπανία. Εξετάζουμε τις συνέπειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στην οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε όμως ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους πολίτες, για την καθημερινότητα των πολιτών και σημαντικά θέματα όπως η απασχόληση, η υγεία, η παιδεία, η, κοινωνική συνοχή, η φτώχεια δεν μπορούν να παραγωνιστούν στον απολογισμό που κάνουμε το έργο της Τρόικα. Ε, δεν μας ενδιαφέρει απλώς ε, η επαναφορά της ε, πίστης ε, της χρηματοπιστωτικής. Τι συνέβη τα τελευταία χρόνια με τα εκατομμύρια των πολιτών που ήταν, έγιναν τα θύματα αυτών των προγραμμάτων διάσωσης, που έγιναν με ραγδαίους ρυθμούς και με τρόπο που προκάλεσε και συγκυριακές ζημίες αλλά και διαρθρωτικές βλάβες. Γιατί όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να έχουν στόχο την ευημερία των πολιτών. Γιατί δεν είναι η Ευρώπη μία λέσχη μόνο πολιτικών προσωπικότητων, αλλά απασχολεί, ανησυχεί για την καθημερινότητα των πολιτών. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτήν την καθημερινότητα, τι συνέβη με τα δικαιώματα των πολιτών, τι συνέβη με την κατάστασή του. Έχουμε εκπροσώπου Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη ε, Ευρω... της, οργάνωσης, Εργασίας και άλλου ε, σημαντικούς ε, καλεσμένους. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαρτίζεται από ε, υπαλλήλους από άνθρωπους, αλλά έχουν, έχουμε ένα ανθρωπιστικό σχέδιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε κηρύγματα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, γιατί έχουμε διεθνή συμβάσει, έχουμε προσυπογράψει τον χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε ευθύνε απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασία. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σα γνώμη, γιατί δεν ζητήθηκε η δική σα γνώμη στη διαβουλεύση. Τι γνώμη έχετε για τι συμφωνίε αυτέ που σύναψε με τι χώρε, ορισμένε χώρε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα μας είπε ότι ε, σε κάποιες στιγμές κρίση θα πρέπει να, ε, να διακινδυνεύουμε ακόμη και θεμελιώδη δικαιώματα. Πού όμως θα πρέπει να μπει το όριο. Γιατί δεν έχουμε μόνο οικονομικές ανάγκες, αλλά έχουμε και άλλες ε, ευθύνες και υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, για να μην επαναληφθούν τέτοιες ε, αντιδράσεις που δεν ήταν ούτε ευρωπαϊκές, ούτε ευφυείς, ούτε λογικές. Και στο μέλλον ε, ε, να διδαχθούμε από τα παθήματα των τελευταίων χρόνων για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη σας σήμερα και την περιμένω με ανυπομονησία γιατί θα ληφθεί υπόψη στην έκθεσή μου που ελπίζω ότι θα τύχει τη ευρεία συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δημιουργήσουμε και πάλι ελπίδες στους συμπολίτες μας. Σε Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σιγητά. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στον Χωσέ Σιλβά Πενέιντα, τον πρώην συνάδελφο που βρίσκεται όμως σήμερα εδώ ως πρόεδρος ε, ε, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Πορτογαλίας και εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, σας είχαμε επισκεφτεί με μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο από το σημερινό, από αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η πατρίδα σας μετά την παρέμβαση της Τρόικα. Θα γίνει λοιπόν ο πρώτος γύρος των παρουσιάσεων. Έχετε 7 λεπτά κύριε Πενέδα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη χαρά επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας εύχομαι καλή χρονιά. Το πρόγραμμα της οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής που διαπραγματευτήκαμε στην Πορτογαλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Απρίλιο του 2011, ξεκίνησε με μια ισχυρή και πολιτική και κοινωνική υποστήριξη. Γύρω στο 80% των βουλευτών της Πορτογαλίας ε, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και μάλιστα είχαμε και ευρεία ε, συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους με την εξαίρεση την Συνομοσπονδία Συνδικάτων σε ZTP-IN. Με στόχο λοιπόν να ε, ε, εφαρμόσουμε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων. Ένα έγκυρο κριτήριο για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματο είναι η σύγκριση των στόχων με τα αποτελέσματα που υλοποιήθηκαν. Σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα, το πρόγραμμα πρόβλεπε για το 2014 μία αύξηση του καθάριστου χώρο προϊόντο στο ΕΠ κατά 2,5%. Η πρόσφατη όμω, που είναι πολύ καλύτερη πρόβλεψη, προβλέπει μείωση μόνο κατά 0,8%. Οι αρχικές προβλέψεις για την ανάπτυξη ήταν τριπλάσιες από τις πρόσφατες προβλέψεις. Η ισορρευτική συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο 2011 με 2013 ήταν γύρω στο 6%. Το Σεπτέμβριο του 2011 το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο υπολόγιζε ποσοστό ενεργείας γύρω στο 14% για το 2013, μία προσωμείωση που τελικά ε, αυξήθηκε σε 17% για τον Νοέμβριο του 2013 και για τον χρόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ε, μια αποκορύφωση της ανεργίας στο 18% για το 2014. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική εξυγίαση, δημόσιο έλλειμμα προβλεπόταν στο 2,3% του ΑΕΠ για το 2014, αλλά τελικά ο σκοπός αυτός, η αρχική αυτή πρόβλεψη διπλασιάστηκε, έφτασε τα 4%. Ε, η εξήγηση για αυτές τις παρεκκλήσεις οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, η ε, παρέμβαση έγινε σε μια χώρα που δεν είχε δικό της νόμισμα και άρα δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κλασικό εργαλείο που συνήθως ε, ισχύει στις παρεμβάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και που είναι η υποτίμηση της ε, χώρας παρέμβασης. Πέραν του καθοριστικού αυτού παράγοντα, το πρόγραμμα διάσωση εξ αρχή ήταν διαποτισμένο από έξι μείζωνα λάθη που οφειλόνται σε μεγάλο βαθμό στην άγνοια τη ε, πορτογαλικής οικονομικής πραγματικότητας. Το πρώτο λάθος ήταν ο ανεπαρκής χαρακτηρισμός της κρίσης και η υποτίμηση της ε, διαρθρωτικής τη διάσταση. Η οικονομική ε, η πορτογαλική οικονομία πάσχει από βασικές ε, διαρθρωτικές ανισορροπίες. Στηρίζεται σε δεκάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έλλειψη κεφαλαίου και τα τελευταία χρόνια σπανίζουν τα κίνητρα για την κατεύθυνση των επενδύσεων σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Δεύτερο λάθος ήταν ε- ότι δεν ελήφθη δεόντως υπόψη η υπερχρέωση των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Τρίτο λάθος, ήταν ότι παραβλέφθηκε το βάρος της εγχώριας ζήτησης και ο τεράστιος αρνητικός αντίκτυπος που είχε η μείωση αυτή της εγχώριας ζήτησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Τέταρτο λάθος. Η αναγγελθήσα μεταρρύθμιση του κράτου ε, δεν έφτασε μέχρι τη δομή τη και έμεινε απλώ σε μια σχεδόν αδιάκριτη μείωση των δαπανών και κυρίω του αριθμού και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τη μείωση των κοινωνικών παροχών και των ε, συντάξεων του, κάτι που επηρέασε το, ε, επηρέασε το εισόδημα των νοικοκυριών και μείωσε κατά πολύ την αγοραστική τους δύναμη. Επίση επιλέχθηκε μια μινιμαλιστική ε, θεώρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της οικονομίας, που ουσιαστικά καταλήξαμε σε μία απλή αλληλουχία εσωτερικών και αντιγωνιστικών υποτιμήσεων και μια δημιουργική, σε μία δημιουργική καταστροφή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ε, ο κοινωνικός αντίκτυπος. Το έκτο λάθος ήταν ε, η έλλειψη χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος. Ως εκ τούτου δεν ελήφθη ε, δεόντως υπόψη ανάγκη προοδευτικής εφαρμογής των μέτρων, αλλά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ε, εφαρμόστηκαν ε, με πολύ απότομο και χονδροειδή τρόπο μέτρα που δεν εξασφάλισαν ελάχιστο ισορροπία και συνοχή των διαφόρων πολιτικών. Πέραν αυτών των έξι λαθών, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Πορτογαλία ξεκίνησε το πρόγραμμα με μια διπλή ανισορροπία. Πέραν αυτών των έξι λαθών, λοιπόν, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Πορτογαλία ξεκίνησε το πρόγραμμα με μια ισχυρή διπλή ανισορροπία. Ε, μια ορατή εσωτερική ανισορροπία με το υψηλό δημόσιο έλλειμμα, το, τη σημαντική ανεργία γύρω στο 9% και μια ισχυρή εξωτερική ανισορροπία γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Σε, επειδή ακριβώ δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε υποτίμηση του νομίσματος, προσπαθήσαμε να διορθώσουμε την εξωτερική ανισορροπία με μια ισχυρή συγκράτηση της εσωτερικής ζήτησης, κάτι που οδήγησε σε μια εκτείναξη στα ύψη της ανεργίας. Γιατί φαίνεται ότι είναι αντιφατική η προσπάθεια διόρθωση ταυτόχρονα της εσωτερική και της εξωτερικής ανισορροπία. Για αυτούς του λόγου, λοιπόν το πρόγραμμα διάσωση τη Πορτογαλίας οδήγησε σε μια διαφορά μεταξύ των στόχων και των αποτελεσμάτων έτσι είχαμε μια πτώση της οικονομικής ε, δραστηριότητας ε, με ιδιαίτερη έμφαση στους ε, δείκτες επένδυσης. Είχαμε μάλιστα μία μείωση 45% μεταξύ του 2009 και 2013 και είχαμε και μείωση της κατανάλωσης. Είχαμε κλείσιμο μεγάλο αριθμό των, επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας, μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών και μία ανεπαρκή δημοσιονομική εξυγίαση. Ε, επίσης είναι ανησυχή η αποδιάρθρωση της ε, κοινωνίας και η εξόντωση ουσιαστικά της ε, μεσαίας τάξης, κάτι που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην λειτουργία μιας, οικονομ... μιας κοινωνικής οικονομίας αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, έχουμε εδώ ένα θέμα που έρχεται σε αντίφαση με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που είναι ακρογωνιαίο του κοινωνικού διαλόγου. Γιατί με βάση τα προγράμματα της Τρόικα και με το επιχείρημα της ανάγκης της μείωσης των του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δημιουργήσαμε προβλήματα στην κανονική διεξαγωγή των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης με, τη δημοσίευση και κάποιων διατάξεων παράτασης, κάτι που δημιούργησε σε απορρίθμιση αγοράς εργασίας. Αυτό το επισήμανε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Είχαμε βέβαια με την πολιτική αυτή και κάποιες θετικέ εξέλιξεις. Μειώθηκε το ε, δημόσιο διαρθωτικό έλλειμμα, κυρίως ε, το πρωτογενές. Και μάλιστα για το 2012 προβλέπεται ένα θετικό υπόλοιπο. Ήδη το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013 αναφάνηκαν κάποια θετικά στοιχεία και φαίνεται ότι είχαμε αύξηση των εισαγωγών σε αντίθεση με την ε, Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία που είχαν πολύ μικρότερη αύξηση των εισαγωγών. Και μάλιστα ε, δυστυχώς τα επιτόκια είναι ακόμη πολύ ψηλά, 5,5% τον Οκτώβριο του 2013, κάτι που φέρνει σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση τις επιχειρήσεις μας. Προσπαθώ με συνοπτικό τρόπο να κάνω μια αξιολόγηση του προγράμματος της Τρόικα στην Πορτογαλία. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε σύστημα προσαρμογής προϋποθέτει οδύνη και θυσίες. Στην περίπτωση όμως της Πορτογαλίας, μια νυφάλια ανάλυση θα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θυσίες και η οδύνη ήταν ε, υπέρ των ε, μεγάλες σε σχέση με τα αποτελέσματα που υλοποίησαμε. Βέβαια, ε, θα ήθελα να πω ότι σας έχω δώσει και ένα παράρτημα μαζί με την ομιλία μου με την γνωμοδότηση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου με μεγάλη συνένεση των κοινωνικών εταίρων και θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών εταίρων προσυπογράφει αυτές τις θέσεις και επίσης θα ήθελα να σας μοιράσω και τη γνωμοδότηση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου μας για την πρόταση προπολογισμού του 2014 που επίσης υιοθετήθηκε χωρίς αντιρρήσεις. Γιατί έτσι δίνουμε το όραμά μας για το μέλλον. Το όραμά μας για το μέλλον στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να έχει και μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Μία δεκαετία και που ταυτόχρονα επιδιώκει τρεις στόχου Την εξηγήση των δημοσίων λογαριασμών αλλά ταυτόχρονα και την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα μια μεταρρύθμιση του κράτου. Είναι σημαντική αυτή η τρει ακρογωνιαίοι λύθοι. Και οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά την παρουσία της Τρόικα, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα και μεγάλη πολιτική συνένεση. Ε, όχι μόνο δηλαδή συνένεση με, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά και μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η θέση και η αξιολόγηση που έγινε από την Πορτογαλία για το έργο της Τρόικα. Euh, euh, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ συγκεκριμένη μαρτυρία για μία από τις χώρες που αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής. Στο πλαίσιο της έκθεσής μας θα δώσω τώρα το λόγο στον Ρέιμοντ Τόρες ως ε, διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ε, είστε γνωστός στα περισσότερα μέλη αυτής της Επιτροπής. Ε, ως υπεύθυνο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είστε πολύ καλόδεχτος να παρουσιάσετε τη μαρτυρία σας εδώ. Όπως ξέρετε πολλοί από εμά. ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι η Τρόικα θα έπρεπε να γίνει ένα κουαρτέτο, να διευρυνθεί ε, Βέβαια, περισσότεροι από εμά θα θεωρούσαμε ότι θα όφιλε να καταργηθεί η Τρόικα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η σχέση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Δυστυχώς, όπως και οι άλλοι, έχετε και εσείς 7 λεπτά για να κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση που απευθύνατε στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική συνάντηση προετοίμασα μία ε, παρουσίαση στα αγγλικά και έτσι θα συνεχίσω στη γλώσσα αυτή. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα προγράμματα οικονομικής βοήθειας σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν ε, περιείχαν ένα μείγμα μακροοικονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όπως ξέρετε, τα προγράμματα αυτά συνοδεύτηκαν ε, με υψηλή και αυξανόμενη ανεργία στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα η ανεργία αυξήθηκε ή παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η αύξηση, και η η αύξηση της ανεργίας και η επιδίνωση της εργασιακής εργασίας ε, είναι μεταξύ των χειρότερων στη σύγχρονη οικονομική ιστορία. Αυτό υπό μία έννοια ήταν αναμενόμενο. Ε, επειδή τα προγράμματα οικονομικής σταθερότητας της Τρόικα συνεπαγόταν, συνεπάγονταν χαμηλότερη ζήτηση. Ε, χαμηλότερη ζήτηση λοιπόν ως ανταπόκριση στις περικοπές ε, σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος. Αυτά τα γεγονότα, οι περικοπές των μισθών και των δαπανών γενικά φυσικά εντείνουν την ανεργία και δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό είναι το κύριο το κυρίως μάθημα που αντλήσαμε. Υπάρχουν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις των προγραμμάτων που εφάρμοσε η Τρόικα και οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις υποτιμήθηκαν στην αρχή. Και υπάρχουν βασικοί λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος βασικός λόγος που είναι γνωστός στους περισσότερους εμπειρογνώμονες της εργασιακής αγοράς είναι ότι υπάρχει μια εγκύτητα μεταξύ... Ε, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Όταν μειώνεται έτσι δραστικά και απότομα η ζήτηση, καταραίουν οι επενδύσεις. Σε όλες τα, τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν αυτά τα προγράμματα, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν άνω του 5%. Σε όλες τις χώρες η, προσ... επενδυτική προσπάθεια είναι πολύ μικρότερη για να ανορθωθεί η οικονομία στις χώρες αυτές. Μιλούμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό μακροπρόθεσμο ε, αποτέλεσμα. Σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απλώς εξαφανίστηκαν. Άλλο ένα σημαντικό μακροπρόθεσμο ε, αποτέλεσμα που εμφανίστηκε βραχυπρόθεσμα όμως και έχει πολλές μακροπροχρόνιες επιπτώσεις γιατί θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ανακάμψουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό. Οι νέοι ε, επηρεάστηκαν δυσανάλογα. Αυτό υπό μία έννοια θα έπρεπε να αναμενόταν γιατί το πρόγραμμα προσαρμογών σήμαινε πολλές περικοπές με λιγότερες θέσεις εργασίας. Ξέρουμε από την έρευνα ότι η ανεργία των νέων, η υψηλή ανεργία των νέων έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις και επηρεάζει όλη τη σταδιοδρομία των ατόμων. Μία άλλη μακροχρόνια επίπτωση είναι η διαδικασία μετανάστευσης από αυτές τις χώρες. Σε όλες τις χώρες όπου έχουμε, από τις οποίες έχουμε στοιχεία, η εξωτερική μετανάστευση διπλασιάστηκε και παραπάνω ίσως τα τελευταία χρόνια από την έναρξη των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικασία αυτή αλλάζει. Τέλος, να αναφέρω τη φτώχεια και τον κίνδυνο φτώχειας. Ε, υπήρχε ένας δείκτης ήταν ένας δείκτης που χρησιμοποιούσε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για πολλές χώρες του κόσμου. Ο δείκτης φτώχειας λοιπόν με την πιθανή εξαίρεση της ε, Πορτογαλίας, όπου ο δείκτης ήταν σχετικός, παρόλο που τελευταίως και στην Πορτογαλία αυξήθηκαν τα ποσοστά φτώχειας. Σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν τέτοια προγράμματα αυξήθηκε ο δείκτης της φτώχειας. Υπάρχει ο δείκτης ε, κατοικίας ε, των μονογονεϊκών ε, οικογενειών. Σε αυτήν την ομάδα του πληθυσμού υπάρχουν διπλά δυσμενή αποτελέσματα για τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών. Ο δεύτερος βασικός λόγος που οι επίπτωσεις ε, των προγραμμάτων αυτών υποτιμήθηκαν ήταν η ασυμμετρία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις συνέβησαν πολύ γρήγορα, ε, μπήκαν βαθιά στην εργασιακή αγορά, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αλλά πολύ λιγότερο και πολύ ανώμια εφαρμόστηκαν σε άλλες αγορές, στα προϊόντα, στα χρηματοπιστωτικό τομέα ή στην ενέργεια. Κατά αποτέλεσμα σε ορισμένες χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και στην Πορτογαλία και σίγουρα και στην Ισπανία, παρόλο που δεν είναι χώρα που εφαρμόζεται πρόγραμμα, παρόλο που ε, μειώθηκαν ε, οι μισθοί και αυξήθηκε η παραγωγικότητα, οι τιμές μειώθηκαν μόνο πολύ σύντομα και δεν αυξήθηκαν τα περιθώρια κέρδους και αυτό ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων υπήρξε πάρα πολύ αργή, ε, πάρα πολύ μερική και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Στην Πορτογαλία ε, δανείζονται με 5,5% ε, ενώ στη Γερμανία με 2% οι χρηματοοικονομικές εταιρείες και πολλές ε, εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση ε, στην ε, τραπεζική πίστη. Λοιπόν, πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό τομέα, στα μέσα κοινωνικής προστασίας, στην εργασία, πολύ ρηχές μεταρρυθμίσεις στους υπόλοιπους τομείς. άλλο τώρα πρόβλημα. Ε, ίσως να θυμόμαστε στη, τη Σουηδία το 1990, τη δεκαετία του 90, η Γερμανία τη δεκαετία του 2000. Υπήρξαν μεταρρυθμίσεις εκεί, αλλά εφαρμόστηκαν σε μια εποχή όπου υπήρχε οικονομική ευημερία, οικονομική πρόεδρος και ήταν, πρόοδος και ήταν εύκολο να προσαρμοστούν οι αγορές αυτές, ιδίως στην Γερμανία, γιατί υπήρχε ανάπτυξη στον κόσμο. Αλλά οι χώρες αυτές που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια πρέπει να αναπτυχθούν σε ένα πλαίσιο που υπάρχει ελάχιστη ανάπτυξη τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Ο άλλος θεμελιώδης λόγος για τον οποίο οι κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας υποτιμήθηκαν ήταν ο σχεδιασμός των ίδιων των μεταρρυθμίσεων της εργασιακής αγοράς. Αυτό, δεν, δυστυχώς δεν έχω χρόνο να επεκταθώ πάνω σε αυτό, να, να δώσω μόνο δύο παραδείγματα. Πρώτον, το θέμα του κανονισμού, των κανόνων απολύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν πολύ γρήγορα με ελάχιστη προσοχή στο σχεδιασμό τους. Σε αντίθεση με την Αυστρία λοιπόν, όπου υπήρξε μια καλοοργανωμένη μεταρρύθμιση σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους που απέφερε πολύ θετικές επιπτώσεις, αυξήθηκε η εσωτερική ευελιξία με διατήρηση όμως των κεκτημένων των εργαζομένων. Στις χώρες για τις οποίες μιλάμε οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν πολύ γρήγορα, μερικές Χωρί χωρίς διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και κατά αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσεις όχι μόνο μείωσαν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, αλλά δεν υποστηρίχθηκαν και οι στόχοι των ίδιων των μεταρρυθμίσεων. Ε, εξακολούθησε να υπάρχει δισκαμψία στην εργασιακή αγορά. Ε, είναι ένα παρόδοξο αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Παρά το βάθος της μεταρρύθμισης δεν επήλθαν τα αποτελέσματα. Και τέλος, φυσικά υπάρχει και εναλλακτική λύση και εναλλακτική τρόπη υπάρχει μια στρατηγική για την ανάπτυξη. Αναφέρθηκε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων. Και τρίτον, πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος εφαρμογής με, μεγαλύτερες, με περισσότερες διαβουλεύσεις. Αν είχαν υπάρξει περισσότερε διαβουλεύσεις, θα ήταν πιο ομαλή η μετάφαση. Ε, και χρειάζεται και συντονισμός. Ελπίζω να έχουμε περισσότερο χρόνο να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά στη συνέχεια τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σα ευχαριστούμε πολύ για τη μαρτυρία σα. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Πέτρο Στάγκο. Είστε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έναν οργανισμό που έπρεπε να αναφέρω όταν ανέφερα και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ένας οργανισμός λοιπόν ο οποίος μέσα στη θεσμική του δομή έχει συντάξει διάφορες γνωμοδοτήσεις για διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των εξελίξεων στην Ελλάδα όσον αφορά ε, σε αυτά που έχουν γίνει και δεν είναι συμβατά με το δίκαιο, έτσι όπως τα έχει εντοπίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένας οργανισμός στον οποίο είναι μέλη όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Ήθελα ευθύ εξ αρχής να πω ότι στη δική μας Επιτροπή δεν συντάσσουμε γνωμοδοτήσεις, συντάσσουμε αποφάσεις και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει στο πλαίσιο της δικής μας Επιτροπής για τα εργασιακά δικαιώματα ως προς την κοινωνική προστασία και την απασχόληση. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων ελέγχει για τη σωστή εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωτών Δικαιωμάτων, την οποία έχουν κυρώσει 47 χώρες μέλη. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μέλη της Χάρτας, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η δική μας Επιτροπή διαχειρίζεται δύο διαφορετικές διαδικασίες. Πρώτον, ετήσιος κύκλος ελέγχου επί τη βάση των εθνικών εκθέσεων που ε, υποβάλλουν οι χώρες μέλη και δεύτερον διαδικασία συλλογική ε, διεκδίκησης, απέτησης αν θέλετε, κάτι το οποίο ε, κάνει την Επιτροπή μας να ανέλθει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενός αν θέλετε δικαιοδοτικού οργάνου, κάτι το οποίο προσωμιάζει την στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το 2003 αποφαθήκαμε λοιπόν επί μια συλλογική διεκδίκηση εναντίον τη Γαλλία με κατηγορία ότι η Γαλλία είχε παραβεί τη χάρτα όποτε η άσκηση ενός από τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη χάρτα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και εξαιρετικά δαπανηρή, κάτι το οποίο ισχύει ε, σε γενικές γραμμές σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης, το κράτος το ενδιαφερόμενο θα πρέπει να φροντίσει να πετύχει τους στόχους της χάρτας σε λογικό χρονοδιάγραμμα με μετρήσιμες επιδόσεις κινητοποιώντας με καλύτερο τρόπο τους σπόρους που διαθέτει και θα πρέπει ε, τα συμβαλόμενα μέρη να ε, μεριμνούν ιδιαιτέρως για τον αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις τους στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στους άλλους ενδιαφερόμενους. Επομένως, τα κράτη τα οποία έχουν προσυπογράψει τη χάρτα και είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόλου δεν έχουν ε, δείξει ε, βούληση να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή της Επιτροπής μας η οποία είναι τόσο ευανάγνωστη και τόσο απλή αν θέλετε και δίνει και περιθώριο ελιγμών. Και υπ' αυτή την έννοια μπορέσαμε να μετριάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία, ε, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα κρατη λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο ετήσιος κύκλος ελέγχου των κρατών επί τη βάση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013 και είναι απογοητευτικός. Απογοητεύουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής που είναι συμβαλόμενοι μέρη στη χάρτα, γιατί ε, ε, δεν προστατεύουν επαρκώς τα συγκεκριμένα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα. Και σας απαριθμώ τη λίστα, τον κατάλογο των άρθρων και των διατάξεων της χάρτας που καταστρατηγήθηκαν και αυτό έχει διαπιστωθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για το δικαίωμα της προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και της συνθήκης υγιεινής στον χώρο εργασίας, δικαίωμα στην κοινωνική αρρωγή, βοήθεια, δικαίωμα των ηλικιωμένων να τύχουν προστασίας έναντι των διακρίσεων, ε, κτλ. λοιπά. Όλα αυτά έχουν καταστρατηγηθεί και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ελέγχου το Δεκέμβριο του 2013 και σημείο αναφορά ήταν η 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2012. Και ε, τα μέτρα που δεν ήταν συμβατά με τη χάρτα βάσει της ε, απόφασης της Επιτροπής μας υιοθετήθηκαν παρατείνοντας κανονιστικούς, ε, κανονιστικές αποφάσεις που επιτάσσουν κοινοτικοί θεσμοί με σκοπό τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να απαλληλθούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Μιλούμε για ε, σύνταξη σε αργότερη, σε μεταγενέστερη ηλικία, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών κοινού, κοινής οφειλίας και το μεταξύ άλλων. Όλα αυτά είναι γνωστά. Στο πλαίσιο λοιπόν της διαδικασίας αυτής της συλλογική διεκδίκησης, αν θέλετε, ε, Επτά φορές εγκαλέστηκε ε, ε, ε, η Ελλάδα και η Επιτροπή εξέτασε και είδε ότι 7 φορές έχουν καταστρατηγηθεί ειδικέ και συγκεκριμένες διατάξεις της χάρτας. Και επομένως η Επιτροπή το 2012 αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβαίνει αυτή τη χάρτα θεσμοθετή ζητώντας ε, βασικό μισθό για τους νέους για την ηλικιακή ομάδα 16-24 που είναι κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Και ε, ε, υπό τις διαταγές της, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν μειώσει την κλίμακα τη μισθολογική στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νέοι Έλληνες και Ιρλανδοί και δημιουργούν έτσι ένα πλαίσιο εργασίας ατυπικό ε, που βγαίνει από το σύνηθες πλαίσιο που έχει να κάνει με την εργασία που παρέχει κανείς, το μισθό που λαμβάνει ή το επίδομα που λαμβάνει όταν είναι άνεργος. Οι χώρες που έχουν δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας μπαίνουν στην εξής κατάσταση. Πρώτον, πρέπει να συμμορφωθούν με νομικές υποχρεώσεις οι οποίες προστασιας μπαινουν στην εξή κατασταση πρωτον πρεπει να συμμορφωθουν με νομικες υποχρεωσεις οι οποιες ειναι αντιφατικές μεταξύ τους και δεύτερον έρχονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση από πολιτική σκοπιάς. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει κανείς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα και τόσο μεγάλη βιασύνη επέβαλε σε χώρες μέλη μέτρα τα οποία τελικά περιορίζουν το επίπεδο προστασίας των ιδιωτών ενώ αυτές οι υποχρεώσεις θα μπορούσε μια χώρα να τις θεωρήσει ασύμβατες με τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει ω χώρα προκειμένου να εφαρμόσει τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, επομένως, ε, η Επιτροπή μας στην απόφαση του 2010 σε σχέση με τις εγκλήσεις έναντι της Γαλλίας για το περιβόητο 35 ώρο, η Επιτροπή μας αποφάθηκε ως εξής δεν είναι στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στο παράγωγο δίκαιο στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι μπορούμε να έχουμε ως τεκμήριο ότι όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβατά με τη χάρτα εξ αρχής. Δεν μπορεί να τεκμέρεται αυτό δηλαδή. Ε, και επομένως έχουμε μειωμένο επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων το οποίο προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδεέστερο του επίπεδου που προβλέπεται από τη χάρτα δικαιωμάτων την οποία έχουν προσυπογράψει τα κρατημέλη και άρα αυτό φέρνει τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δύσκολη θέση νομική, πολιτική και μια θέση αντιφατική. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ε, κατά πόσο το εργασιακό δίκαιο της Ένωσης συνάδει με τη χάρτα, γιατί η Ένωση δεν είναι μέλος της χάρτας. Οι χώρες μέλη είναι. Από την άλλη πλευρά, η νομολογία της Επιτροπής μας από το 2010 μέχρι σήμερα ε, λέει ότι οι υποχρεώσεις στα συμβαλόμενα μέλη, δηλαδή στις χώρες που έχουν προσυπογράψει τη χάρτα, οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα απαλλάσσουν τα κράτη-μέλη από την υποχρέωση τους επίσης να εφαρμόσουν σωστά τη χάρτα αυτή και οφείλουν στη δική τους ένωμη τάξη να προβλέψουν και να μεριμνήσουν ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της χάρτας. Επομένως, από τον Ιανουάριο του 2013, εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νομική προστασία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ένωσης, ειδικότερα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Και κάνουμε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Δικαστήριο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ως Επιτροπή ότι η Ένωση χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα, διότι έτσι θα έχει ένα σεωρευτικό αποτέλεσμα που θα είναι πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Σημείο αναφοράς δεν θα είναι μόνο η αγορά ε, και οι αγορές, αλλά και τα ε, υποκείμενα δικαίου έτσι όπως ε, τα αντιλαμβάνεται και τα ερμηνεύει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και η δική μας Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την συμπληρωματική αυτή παρουσίαση. Θα δώσω τώρα το λόγο πάντοτε για 7 λεπτά στον τελευταίο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τόχσεν Σούλτεν είσαστε επικεφαλής ε, του τμήματος ε, πολιτικής και μισθών ε, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, στο Γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSE και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα. Υπήρξε ε, μέλος του Συμβουλίου G και του Ιδρύματος Hans Wöttler. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ καταρχήν θερμά για την πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Ινστιτούτου μας, αλλά και άλλων Ινστιτούτων, γιατί πρόκειται για ένα δίκτυο διαφορετικών Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων από 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα μερικά από τα Ινστιτούτα αυτά βρίσκονται σε χώρες τις οποίες αναφερθήκαμε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ε, μία βασική πτυχή, στις ε, συνέπειες της πολιτική τη Τρόικα στους μισθούς, αλλά και στο γενικό σύστημα των μισθών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό θα είναι το κεντρικό στοιχείο της παρουσίασής μου. Φυσικά, ε, στόχος της Τρόικα ήταν ε, να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών και θεώρησαν ότι θα το επιτύχουν αυτό με μείωση του κόστους εργασίας. Και γι' αυτό εφάρμοσαν δύο ε, στρατηγικές, μία άμεση παρέμβαση στις, ε, στην εξέλιξη των μισθών και κυρίως περικοπές στους μισθούς και πάγωμα στους μισθούς και η δεύτερη μέθοδος ήταν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με επεμβάση τον τρόπο σύναψης των συλλογικών ε, συμβάσεων. Ε, η πρώτη μέθοδος ήταν η άμεση παρέμβαση στην ίδια την πολιτική των μισθών με περικοπές κυρίως και παγώματα μισθών. Είδατε ε, από διάφορα έγγραφα όλα τα στοιχεία, δεν θα τα επαναλάβω, είδαμε μειώσεις στις τάξεις 30, 40 έως και 50% των μισθών στο δημόσιο. Τουλάχιστον ε, στις ε, τέσσερις χώρες που εφάρμοσαν προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Επίσης είδαμε μείωση του κόστους, μείωση ακόμη και του κατώτατου μισθού ή πάγωμα μισθών. Είχαμε σημαντικές τέτοιες μειώσεις στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία είχαμε μειώσεις των μισθών με απότερο σκοπό βέβαια να μειωθούν οι απολύσεις και να γίνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερες οικονομίες. Αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό και που δεν εμφανίζεται συχνά, δεν ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ήταν οι συνέπειες της παρέμβαση της Τρόικας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικέ συμβάσεις. Γιατί οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας επηρέασαν και τις ε, συλλογικέ διαπραγματεύσεις και συμβάσεις. Βέβαια, μερικές φορές ε, διερωτόμαστε ποια θα ήταν η ε, ιδανική συλλογική διαπραγμάτευση και η ιδεώδης συλλογική σύμβαση. Οι κοινωνικοί εταίροι, ε, ή μάλλον η Τρόικα τροικα τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης ε, του, του, της κάλυψης της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ε, μείωση του εύρους των συμφωνιών, μία αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ένα τρόπο λιγότερο κεντρικό για τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης έχουμε στην έκθεση τη μείωση των μισθών και τη μείωση της επιρροής των συνδικάτων στον καθορισμό των μισθών. Ενώ ταυτόχρονα είχαμε μείωση ή περιορισμό της αρχής ευνικότερης ρύθμισης. Τι τι συνέβη λοιπόν με την παρέμβαση της Τρόικας ε, επιβάλλει όλες αυτές τις ε, υποχρεώσεις, όλες αυτές τις συστάσεις που γίνονται δεκτές ε, σε εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είχαμε δύο ή τρεις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις αγοράς εργασίας με την αρχή της ε, κατάργησης της ευνοϊκότερης ρύθμισης ή της ε, απέτησης της ε, απόδοσης, της μεγαλύτερης απόδοσης και βλέπουμε ότι στις χώρες της διάσωσης έχουμε μια ορατή υποχώρηση των τομεακών συλλογικών συμβάσεων και μεγαλύτερη έμφαση στις συμβάσεις που γίνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων και που υπερέχουν των τομεακών συμβάσεων. Και στο 80% των περιπτώσεων είχαμε καθορισμό των κατώτερων μισθών σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που πρόβλεπαν οι συλλογικές συμβάσεις. Στις ε, χώρες ε, της διάσωσης που σε, μεγάλες, σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις α, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαμε πολύ αρνητικές συνέπειες για αυτές. Και στη, στην Πορτογαλία αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Βλέπουμε στην Πορτογαλία 1,2 εκατομμύρια ε, των εργαζομένων που υπόκεινται σε συλλογικές συμβάσεις και το 2011 και το 2012 είχαμε 328.000, δηλαδή από 1,2 εκατομμύρια περάσαμε στους 328.000 ε, κάλυψη. Τεράστια μείωση της κάλυψης δηλαδή των εργαζομένων από τις συλλογικέ ε, συμβάσεις. Οπότε δεν είχαμε πια οικουμενική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης άλλαξαν τα κλασικά συστήματα ε, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνικής εταιρικής σχέσης. Στην Κύπρο Είχαμε ένα ήδη αρκετά αποκεντρωμένο σύστημα και εκεί ε, επικεντρώθηκα σε τη μαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Προσπάθησαν δηλαδή να αναχαιτήσουν αυτήν την αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Η Ισπανία δεν εφάρμοσε πρόγραμμα διάσωσης, αλλά υπογράφηκε παρόλα αυτά ένα μνημόνιο, μνημόνιο συνεννόησης και στο μνημόνιο αυτό απαιτήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις και από την Ισπανία και μάλιστα έγινε μια ριζοσπαστική μεταρρυθμίση στην οποία περιορίστηκε η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων. Δεν υπάρχει πια υποχρεωτικός χαρακτήρας των συλλογικών συμβάσεων. Την τελευταία τετραετία διαπιστώσαμε ότι η πλειοψηφία των χωρών μείωσαν τους μισθούς τους ε, και έτσι μειώθηκε κατά πολύ το εργασιακό κόστος. Και έρχομαι στα συμπεράσματα μου. Η Τρόικα κάτι που δεν αναγνωρίζεται συχνά, προώθησε ρήξη και έλευθες και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις ε, παντού στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων. Αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων, τεράστια παλινδρόμηση της ίδιας της έννοιας της συλλογική σύμβασης ό,τι αφορά την κάλυψη. Περιορίστηκε δραματικά η κάλυψη και δημιουργήθηκε μια τεράστια υποτίμηση, απαξίωση των ε, συλλογικών συμβάσεων. Και επίσης υπήρχε μια μεγάλη πίεση των μισθών προς τα κάτω. Ένα σπιράλ αποπληθωριστικό με πολύ ε, δυσμενείς συνέπειες στην ζήτηση και στην αγοραστική δύναμη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους τέσσερις εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι μας παρουσιάσατε απόψεις εξαιρετικά διαφωτιστικές, οι οποίες συμπλήρωναν η μία την άλλη. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους εμπειρογνωμοσύνη για να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της παρέμβασης της Τρόικας στις τέσσερις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους σκιώτες εισηγητές μου έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Ρεζίνα Ντεμπάστος. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. οι νέες σημειώνω για να οργανώσω καλύτερα τη συζήτησή μας και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, για να οργανώσουμε καλύτερα τις εργασίες μας, σας προτείνω λοιπόν τρία λεπτά να έχει ο κάθε σκιώδης εισηγητής στη διάθεσή του και δύο λεπτά να έχει κάθε μέλος της Επιτροπής μας για να ε, θέσει ερώτηση ή να κάνει σχόλιο. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο. Ρεζίνα Μπάστος, είναι Τσουμπόρ, Άννα Γκόμες, Τόμας Μαν, Χατζηγεωργίου, Σοφοκλέους, Κοστέλο, Εστρέλα και βεβαίως ο εισηγητής. Ξέχασα κάποιον. όρι Πενάρα, Μπάτο. Αυτά. Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος των παρεμβαίνοντων. Ρεζίνα Μπάστος, λοιπόν, τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους τέσσερις εμπειρογνώμονές μας που μας εξήγησαν ε, τις απόψεις τους ε, για το τι πάει στραβά στα προγράμματα διάσωσης των τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τεσσάρων χωρών δηλαδή που δέχτηκαν την οικονομική ενίσχυση της Τρόικας και υπευλήθησαν σε προγράμματα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο κύριος Σέρκας που είναι συγητής ε, της ε, Επιτροπής μας θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου της Τρόικας στις τέσσερις αυτές χώρες και ε, θα κάνουμε πρώτα απ' όλα μια σωστή πλαισίωση, που η πλαισίωση είναι διαφοροποιημένη ανάλογα με τη χώρα, γιατί οι αιτίε που οδήγησαν την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία στο να αποτανθούν στην Τρόικα είναι διαφορετικέ. Όλε όμω οι αιτίε και όλοι αυτοί οι λόγοι είναι πολύ σοβαροί. Στην πατρίδα μου, την Πορτογαλία, μετά την σοσιαλιστική διακυβέρνηση δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δημόσιο χρέο ένα πολύ ευάλωτο δημόσιο χρέος και ένα δημόσιο έλλειμμα που ε, άφησε ε, σαφή μια κατάσταση της Πορτογαλίας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Γι' αυτό και χρειάστηκε να αποτανθεί στην ε, Τρόικα και να ζητήσει δάνειο 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν ελάβανε αυτό το δάνειο δεν θα μπορούσε το, το κράτος να πληρώσει τι υποχρεώσει του ούτε σε επίπεδο μισθών, ούτε σε επίπεδο συντάξεων, ούτε να αποπληρώσει το χρέος του, ούτε να χρηματοδοτήσει τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και το πλαίσιο είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα. Βέβαια, συμφωνούμε ότι το πρόγραμμα διάσωσης που εφαρμόστηκε είχε σε όλες τις χώρες τεράστιες κοινωνικές συνέπειες κοινωνικές συνέπειες σε επίπεδο ανεργίας. Είχαμε αύξηση της ανεργίας ανδρών, γυναικών και νέων στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία. Πολύ ανησυχητικά τα επίπεδα ανεργίας. Παρόλο που στην Πορτογαλία τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε μια πολύ θετική μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, αλλά και του γενικού ποστού της ενέργειας και είχαμε κάποια ε, θετικά, θετικά δείγματα της οικονομίας. Πάντως το πρωταρχικό λάθος ε, που επισήμανε ο συνάδελφος Πενέδα, τον οποίο καλωσορίζω εδώ, στο σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος διάσωσης ε, στην Πορτογαλία, ήταν ο ελάχιστος χρόνος που αφιερώθηκε στην εκτέλεση του προγράμματος. Είναι αναφισβήτητο ότι μία τριετία για την εκτέλεση ενός προγράμματος που έχει τόσο τεράστιες διαρθρωτικές ε, πτυχές και συνέπειες και μεταρρύθμισε χρηματοπιστωτικό, κοινωνικό, οικονομικό τομέα, έχει ένα τεράστιο τίμημα αυτός ο ελάχιστος χρόνος και είναι σαφές το τίμημα που καταβάλαμε. Είναι ορατό, είναι αδιαφυσβήτητες πια οι αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που έχει αυτό το τίμημα για τους πολίτες. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής ποια είναι τα μέτρα, ποιοι είναι οι φορείς, ποιος είναι ο τρόπος δράσης ε, που θα, που θα προσφέρει στο μέλλον ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που επαναληφθεί μια τέτοια κρίση, κάτι που φυσικά το απευχόμαστε. Αυτό είναι το θέμα, γιατί το ζήτημα της πίσης του χρόνου και το ελάχιστο χρόνο που είχαμε για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ήταν σαφές. Και μάλιστα το αναγνώρισε και η, Διευθύντρια του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου. Και οι εμπειρογνώμονες που ε, αξιολόγησαν ε, την εκτέλεση του προγράμματος δυστυχώς ήταν ανελαστική, αδιάλακτη και δεν ε, συμφώνησαν σε καμία παράταση χρόνου προς τις χώρες για να εφαρμόσουν τα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να στιγματίσουμε, να στυλιτεύσουμε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που δόθηκε για την εκτέλεση τόσο σημαντικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζουμπέρ και να σας υπογραμμίσω ότι έχουμε εδώ μια δημόσια ακρόαση. Οπότε καλό θα ήταν να θέτετε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες, να αξιοποιήσουμε την παρουσία τους και να εμβαθύνουμε περισσότερο στα θέματα. Είναι σε Ζούμπερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ και να στο θερμά τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Πενέτα Σίλβα και να θέσω μερικές ερωτήσεις. Από αυτά που άκουσα, διαπίστωσα ότι η διάγνωση για την αξιολόγηση του έργου της Τρόικα συμπίπτει με τη διάγνωση που έκανε το δικό μου κόμμα για το έργο της Τρόικα. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που διαγνώστηκαν λάθη, τόσο σοβαρά που διακύβευσαν και την ίδια την οικονομική ανάπτυξη των χωρών διάσωσης. Γιατί δεν αντιστράφηκαν, γιατί δεν τροποποιήθηκαν ριζικά αυτά τα μέτρα. Το θέμα της ε, εσωτερικής ζήτησης αναδειχθήκε ως μείζον πρόβλημα ε, των χωρών που εμπόδισε την οικονομική ανάπτυξη. Αν όντως συρρυκνώθηκε αυτή η εσωτερική ζήτηση, γιατί δεν αυξήθηκαν οι μισθοί, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν οι μισθοί, γιατί δεν ε, αναβαθμίστηκαν οι συντάξεις, γιατί δεν ενισχύθηκαν τα κοινωνικά επιδόματα, γιατί δεν αναβαθμίστηκε η συλλογική διαπραγμάτευση, ώστε να μην επιτραπεί η μείωση των μισθών. Δεν έπρεπε αυτά τα μέτρα να ληφθούν αν θέλαμε πραγματικά να ενισχύσουμε την εσωτερική ζήτηση και να τονώσουμε την οικονομία αυτών των χωρών. Ενώ το αντίθετο τελικά συνέβη με τα μέτρα και τη λογική ε, του, του προγράμματος ε, της Τρόικα. Εμείς ε, ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Συνεπειών ε, εξετάζουμε τις κοινωνικές συνέπειες των μέτρων, αλλά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πλήρως τις κοινωνικές συνέπειες από τις οικονομικές, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το οικονομικό με το κοινωνικό σκέλος. Τα μέτρα της Τρόικα οδήγησαν σε φτώχεια, εξαθλίωση και αύξηση της αποδημίας από τις χώρες διάσωσης, ενώ ταυτόχρονα ε, αύξησε αστρονομικά τα κέρδη των πολυεθνικών και των ε, πολυεκατομμυριούχων. Αυτά ήταν τα στρεβλά ε, αποτελέσματα των ε, δραστηριοτήτων και της εφαρμογής του προγράμματος. Έχω και ένα άλλο ερώτημα. Αναφέρθηκε ότι τα επιτόκια που πληρώνουν οι χώρες αυτές είναι ανυπόφορα, είναι αβάστακτα. Και με τα υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη. Με τέτοια χρέη και με τέτοια επιτόκια πώς θα επιβιώσουν αυτές οι χώρες. Γιατί ήδη ε, υπάρχει ύφεση, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Οπότε είναι αδύνατο να πληρώσουν με τόσο υψηλά επιτόκια μέσω και πρόθεσμα τα χρέη τους αυτές οι χώρες. Οπότε δεν θα ήταν καλύτερη λύση μια αναδιαπραγμάτευση του χρέους πέραν άλλων μέτρων που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ είμαι και οδησηγήτρια της ομάδας μου, της ΓΚΟΕ, για την έκθεση αυτή και η θέση μας από την αρχή ήταν κατά της ύπαρξης της Τρόικα και σε καμία περίπτωση δεν θα δώσουμε την συμφωνία μας σε μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στην Άννα Γκόμες για δύο λεπτά. Um, Um, Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, συμπατριώτη μου και όπως είπε και εκείνος, οι, οι θέσεις του αντανακλούν τις απόψεις των συνδικάτων και των εργοδοτικών οργανώσεων. Υπήρξε μια αντιπροσωπεία που πήγε πρόσφατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισαβόνα και τα τσέκαρε όλα αυτά. Υπήρχε, μιλήσαμε για την περίπτωση ενός ατόμου που πέθανε από καρκίνο γιατί δεν μπόρεσε να κάνει ορθοσκόπηση όταν χρειάστηκε. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν τρόφιμα για φάρμακα. Υπάρχουν παιδιά που πεινάνε ε, και τρώνε μόνο στο σχολείο. Ε, η ανεργία, ναι, έχει λίγο μειωθεί, αλλά η ανεργία των νέων αυξάνεται. Στο 37% μάλιστα πάνω από 200.000 ε, των πλέον προσοντούχων ατόμων έχουν φύγει από τη χώρα. Πρόκειται για το πιο αποτρόπαιο πλήγμα ε, στην ε, πιθανότητες βιωσιμότητας της οικονομίας της Πορτογαλίας λόγω των πολιτικών που έχει επιβάλει η Τρόικα. Η κυβέρνηση απορρίπτει, προσπαθήσει να, προσπαθεί να καταργήσει τη συνταγματική, την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου σχετικά με τις ε, συντάξεις και τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Ε, υπάρχουν οι δυτικοποίησεις, παρόλο που δεν ε, περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται. καμία από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που μας υποσχέθηκαν δεν πραγματοποιούνται και ιδίω οι μεταρρυθμίσει που έχουν να κάνουν με την περικοπή των υπέροχων κερδών των επιχειρήσεων, ε, των μεγάλων επιχειρήσεων. Ε, λόγω των υπευθύνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου, του κοινωνικού χάρτη και των κοινωνικών δικαιωμάτων, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το δημοκρατικό έλεγχο για το μέλλον. Η Επιτροπή αυτό που μπορεί να κάνει ε, και το Κοινοβούλιο και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να είναι όπως είναι, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικές παραμέτρους και τους μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, όχι μόνο για τη δική μου χώρα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη και την οικονομία. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος. <clears throat> Äh, Θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Αλεχάνδρο. Προφανώς και εξετάζουμε τον λόγο, εξετάζουμε την ευθύνη των ατόμων ε, της ελίτ. Ε, θέλουμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι κάποια μέτρα είναι απαραίτητα. Φυσικά και πρέπει να υπάρξει τακτοποίηση των προϋπολογισμών και των οικονομικών. Εκείνα τα άτομα που δεν κατέβαλαν φόρους πρέπει φυσικά να υποχρεωθούν να τους καταβάλουν. Ε, ε εντάξει, η Τρόικα δεν είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Βελζεβούλ, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν συναποφασιστεί από όλες τις πλευρές ε, και πρέπει τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και ότι οι, ρυθμίσεις αυτέ οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα αποβούν ευνοϊκές και θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και μεγέθυνση. Μιλάτε για συμμετρία ή μάλλον για έλλειψη συμμετρίας. Χρειαζόμαστε, λέτε, μεταρρυθμίσεις, αλλά όχι να τις επιβάλλουμε ταχύρυθμα. Ε, εάν ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές σε ένα πιο μεγάλο χρονικό πλαίσιο, τότε σίγουρα θα μπορέσουν οι άνθρωποι να προσαρμοστούν κτλ. Δεν μπορούμε όμως να σταματήσουμε αυτό που έχει ξεκινήσει, γιατί τα, χρειαζόμαστε αυτά τα μέτρα. Ίσως βέβαια να ήταν πιο αποδεκτά εάν μπορούσαμε να τα εφαρμόσουμε σε μακρύτερο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τις ε, ευκαιρίες της Τρόικα ότι έχουν γίνει κάποιες επιτυχίες. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι βελτιώθηκε η λογοδεσία. Βέβαια χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευθύνη και πρέπει η Τρόικα να υποβληθεί σε λογοδοσία. Πρέπει όμως όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές και έχει συμβεί. Αν δείτε την Ιρλανδία, ε, η Ιρλανδία έχει βγει από την ομπρέλα, ε, ε, από την της Τρόικα. Και η Ισπανία είναι χωρίς μνημόνιο αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Κύριος, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν έχω καμιά πίστη ότι θα βγει οτιδήποτε από αυτή μας τη συνεδρία. Λυπούμε που ακούγουμε απεσιόδοξος. Έχω συμμετάσχει και σε άλλες συνεδρίες. Είμαστε λίγο του μπλα μπλα. Το Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας να έχει ουσιαστικό ρόλο. Και αν δεν κατακτηθεί αυτό, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικό. Το, το δεύτερο που έχω να πω έχει πει ο κύριος ε, Σέρκας προηγουμένως, ε, ελπίζω να προφέρω καλά το όνομά του, ότι πρέπει να αποδείξουμε, είπε, ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και το ανθρωπιστικό στοιχείο στις συνεδριάσεις. Δεν αναφέρομαι τώρα στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, αλλά στις συνεδριάσεις της Τρόικα που παίρνει τις αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει ο ανθρωπισμός, αγαπητέ μου φίλε, διότι ένας άνθρωπος που παίρνει 20.000 ευρώ το μήνα 40 ίσως φορές περισσότερα λεφτά από όσα παίρνει ο μέσος εργαζόμενος στις χώρες που είναι στο μνημόνιο. Ο άλλος παίρνει 500 ευρώ και εσύ παίρνει 20, όταν λέω εσύ αναφέρομαι στους ανθρώπους της Τρόικα, δεν μπορεί να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι θες κάνει. Δεν μπορεί να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα είδος υπερανθρώπου. Έχει μια πανοπλία των 20 και πλέον χιλιάδων ευρώ τον, τον μήνα. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο, δεν θα αναφερθώ στα νούμερα και τα στοιχεία, την υπερβολική αύξηση της ανεργίας, το τι συμβαίνει με τον κόσμο και τις ουρέσεις στα νοσοκομεία, με τα παιδιά στο σχολείο που λιποθυμούν επειδή δεν έχουν ένα ποτήρι γάλα. Δεν θα τα πω αυτό για να μην δείξω ε, έλλειψη κουράγιου ε, από τον κυπριακό λαό. Αλλά θα πω το εξή. Τα προβλήματα στην Κύπρο ήρθαν επειδή η χώρα μπήκε στο ευρώ. Και μετά ήρθαν αυτοί που υποχρεωτικά μας έβαλαν στο ευρώ να λύσουν τα προβλήματα με τον τρόπο Merci, cher collègue. Je donne maintenant la parole à Monsieur Sophocleus. Διακόπτη η πρόεδρος. Ε, θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο που σας έχω δώσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σοφοκλή. Τα μέτρα που πήρε ή απέτησε όχι μόνο δεν έφεραν αποτελέσματα, αλλά ενίσχυσαν ακόμη περισσότερον την ύφεση και την ανεργία. Αποδιοργάνωσαν των κοινωνικών ιστών των κρατών. Ενίσχυσαν δυστυχώς την αφισβήτηση των πολιτών κατά της Τρόικας και βέβαια κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ενδιαφέρον τους εξαντλήθηκε στους αριθμούς και όχι στους ανθρώπους στις τιμές των αγαθών και όχι στην πραγματική τους αξία για να θυμηθούμε λίγο τον νομπελίστα τον Κρούκο. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ελλάδα, ανεργία 27,4%, όρια της στόχιας 31%. Κύπρος 17,8%, όρια της στόχιας 25%. Πορτογαλία 15,5%, όρια της στόχιας περίπου 25%. Ιρλανδία 12,3%, όρια της στόχιας 29,4%. Τουλάχιστον εδώ και τώρα ας παραδεχτούν πρώτα και πάνω απ' όλα είναι καθήκον τους τα λάθη τα οποία έχουν κάνει. Αλλά ταυτόχρονα και το δεύτερο είναι πιο σημαντικό είναι η αλλαγή αυτής της αντιπαραγωγικής πολιτικής. Η οικονομία αγαπητοί συνάδελφοι θέλει επενδύσεις, θέλει έργα, θέλει φρέσκο χρήμα θέλει θέσεις νέες εργασίας. Αυτή μπορεί να είναι η λύση. Και όχι η λιτότητα και τα ληστρικά μέτρα. Επιτέλους, ας το κατανοήσουν ή καλύτερα, ας το κατανοήσουμε. Ευχαριστώ. Διαπιστώνω ότι πολύ λίγοι θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονές μας. Είμαστε σε ένα πλαίσιο ακρόασης τεσσάρων εμπειρογνωμόνων που έχουν πράγματι ε, τη δυνατότητα να μας διαφωτίσουν. Η Ελίζα θα έχει το λόγο για δύο λεπτά και μετά ο κύριος Κοστέλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων και κυρίως την παρουσίαση του πρώην συναδέλφου, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε μακρόν ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή μαζί σας και με ενδιαφέρει, ε, θεώρησα πολύ ενδιαφέρουσα και οφείλω να το ομολογήσω αυτό, ε, την κριτική σας, την αξιολόγησή σας. Με πολύ εύγλωτο τρόπο υπογραμμίσατε τα κενά και τα λάθη στα προγράμματα που εφαρμόζει η Τρόικα στις χώρες μέλη. Είναι κάτι που ασφαλώς μας ανησυχεί όλους εμάς ως Επιτροπή. Ε, κοινοβουλευτική και οφείλουμε να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτό το οποίο κάνει η Τρόικα, να συνεργαστούμε με τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, ούτως ώστε κάθε φορά που προτείνεται μία μεταρρύθμιση να είναι ευφυής, να είναι έξυπνη, να είναι χρήσιμη για τον τοπικό πληθυσμό. Μιλούμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πράγματι θα μπορούσαν να είχαν γίνει και να έχουν γίνει ήδη, να μην μείνουμε στην επιφάνεια. Αυτό έχει άλλωστε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό και είναι κάτι που πρέπει να πούμε. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε πολύ καλά το κοινοβούλιο μας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία με τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, εμείς ως Επιτροπή Κοινοβουλευτική, ως Κοινοβούλιο, για να αποφύγουμε λάθη της Τρόικας στο μέλλον και να μπορέσουν να συγκροτηθούν οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κοστέλο και μετά η κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θέρκας και τους εμπειρογνώμονες για την παρέμβασή τους. Οι παρουσιάσεις τους ήταν εξαιρετικά χρήσιμες. Είναι ευρία η συνένεση. Πολλά λάθη έχουν γίνει από την Τρόικα. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω ότι παρόλο που ξεφύγαμε από την Τρόικα, η κληρονομιά της θα μας τυχιώνει για πολλά χρόνια ακόμα. Ερωτώ λοιπόν, Είδαμε και ακούσαμε σήμερα στην ακρόαση ότι η Τρόικα έκανε λάθη και αυτό είναι γεγονός. Παρόλα αυτά είναι ευρεία η βούληση να συνεχιστεί η πολιτική της λιτότητας, της δημοσιονομικής αυστηρότητας. Η Ιρλανδία απόλεσε την οικονομική της εθνική κυριαρχία το Δεκέμβριο του 2010 και την αποκατέστασε τον ε, περασμένο Δεκέμβριο, πριν από ένα μήνα, αλλά με πολύ μεγάλο κόστος κοινωνικό, εργασιακό. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε θέματα κοινωνικής προστασίας, δημοσίων υπηρεσιών, τεράστιος αντίκτυπος ε, στην ανεργία, μετανάστευση προς το εξωτερικό είναι και ειδικότερα των νέων. Χάσαμε το 1 τέταρτο της νεολαίας μας. 176.000 νέοι από το 2009 μέχρι σήμερα έφυγαν στο εξωτερικό και αν δεν καταφέρουμε να προσελκύσουμε και να έχουμε ε, εργασιακό δυναμικό ε, με μεγάλη κατάρτιση, τότε δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης υψηλού επίπεδου στο μέλλον. Έρχονται τα μέλη της Τρόικας και ασχολούνται ε, με τη διαβούλευση, αλλά είναι μια ψεύδοδιαβούλευση. διαβούλευση. Έλεγαν ότι θα διαβουλευθούν με δικαλιστές, με όλους τους φορείς της κοινωνίας, όμως τελικά ο αντίκτυπος το feedback που είχαμε από τους συνομιλητές τους ήταν ε, ε, διαφορετικό. Ε, και ξέρετε, πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ουσιαστικέ προτάσεις για επενδύσεις, για ανάπτυξη, για δημιουργία θέσης απασχόλησης. Τις έχουν ε, υποβάλει επανειλημμένως και η Τρόικα πάντοτε το να ακούσει, χωρίς να έχει οποιαδήποτε δημοκρατική νομοποίηση. Ερωτώ, πώς μπορεί να γίνει η Τρόικα πιο υπόλογη από τη δημοκρατική σκοπιά. Ποιος είναι ο τρόπος να αρχίσει ε, να αναφέρει και να αποδοθεί λογαριασμό. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά Κυρία Δίτα Στρέλα, θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα τον εισηγητή μας, τον Αλεχάνδρο Σέρκας, για την αξιοθαύμαστη δουλειά του. Να ευχαριστήσω ε, και τους ε, εμπειρογνώμονές μας, ιδιαίτερα τον συμπατριώτη μου τον κύριο Πενέντα και να περιοριστώ σε κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται προς τον ε, κύριο Σίλβα Πενέντα δεδομένη της διάγνωση που έκανε για την κατάσταση της ε, πορτογαλικής οικονομίας και την συστηματική διαφορά που διαπιστώσαμε μεταξύ των προβλέψεων και των αποτελεσμάτων ε, και με την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης ε, στην Πορτογαλία και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάιο θα τερματιστεί το πρόγραμμα προσαρμογής, δημοσιονομικής προσαρμογής και θα εξέλθει από αυτό η Πορτογαλία. Αυτό θα σημάνει το τέλος της λιτότητας, ε, θα σημάνει τη μείωση των επιτοκίων και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πορτογαλικής οικονομίας. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα προσαρμογής, το χρέος των ιδιωτών, των οικοκυριών στην ε, Πορτογαλία ήταν το διπλάσιο του δημόσιου χρέους. Τι συνέπειες ε, είχε αυτή η διαφορά στην ε, επιδείνωση της κατάστασης των οικοκυριών, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο δημόσιο χρέος που ήταν υψηλότερο, το 90% του ΕΚ, σήμερα όμως είναι περίπου 130% του ΕΠ. Οπότε και το δημόσιο χρέος ε, ε, μεγάλωσε παρά την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής. Οπότε αυτές τις ερωτήσεις έχω προς τους εμπειρογνώμονές μας. Και δεδομένου ότι πολλοί οικονομολόγοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και μάλιστα ακόμη και βραβεία Νόμπελ Οικονομίας έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου κατά των αρνητικών συνεπειών αυτής της υπερβολικής δόσης λιτότητας. Γιατί λοιπόν δεν εισακούστηκαν οι φωνές και οι τους από τις εθνικές αρχές ή τις ευρωπαϊκές αρχές, από τους ηθήνοντες, γιατί θα θα πληρώσουν ε, οι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης τις αρνητικές συνέπειες που επέφεραν στους πολίτες. Παρακαλώ, ήδη έχουμε μισή ώρα καθυστέρηση, γνωρίζω ότι είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό το θέμα, αλλά έχουμε πολλούς ε, εγγεγραμμένους στον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Τσάμπα Όρη και μετά η κυρία Μπεναμπάρ Αντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά και με ζωηρό ενδιαφέρον τις ομιλίες των εμπειρογνωμόνων και θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για την πατρίδα μου, την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία ήταν από τις πρώτες χώρες που βρέθηκαν στο χείλο του γκρεμού, στο χείλο της χρεοκοπίας. Και ζήτησε συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήψε και δάνεια με διεθνείς οργανισμούς. Κάτι που μας βοήθησε τελικά με αυστηρά μέτρα λιτότητες να διορθώσουμε την κατάσταση. Βέβαια, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επανεκλέγει και η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε την ίδια κατάσταση. Έχουμε πολλές πολυεθνικές και πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς και τράπεζες που συμμετείχαν στην διαδικασία που ξεκίνησε στην Ουγγαρία. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, πολλά τα διευθετήσαμε και με πολύ κόπο και προσπάθεια καταφέραμε να αποπληρώσουμε το χρέος προς την Παγκόσμια Τράπεζα που ήταν κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Καταφέραμε τελικά να επιτύχουμε και 1% οικονομική ανάπτυξη το τελευταίο χρόνο. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς και εκεί διαπιστώνουμε μία ανωδική πορεία. Εμείς λοιπόν στην Ουγγαρία ακολουθήσαμε τελείως διαφορετική μέθοδο και κατεύθυνση. Και προσπαθήσαμε με διάφορα μέτρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τώρα δρεύουμε τους καρπούς αυτής της στρατηγικής. Τι γνώμη έχουν οι εμπειρογνώμονες. Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και αξίζει να διερευνήσουμε και εναλλακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεναμπάρ Ατού για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι πλήρως ε, τις αναλύσεις και τη θέση του εισηγητού μας του κύριου Σέρκας ακούγοντας για τις ζημίες που προκάλεσαν τα μέτρα της Τρόικα, ε, σκέφτομαι το σχέδιο ε, διαρθρωτικής προσαρμογής που εφαρμόσαμε για τις ε, φτωχέ χώρες. Τελικά, οι ίδιε αιτίε οδηγούν στις ίδιες συνέπειες, δηλαδή καταστροφή της κοινωνικής προστασίας, αποδυνάμωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, παταγώδης αποτυχία της Τρόικα, που είναι και αναφυσβήτητη. Οι συμπολίτε μας λοιπόν βλέπουν την κατάσταση και θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν τους βοηθάει και εκεί το πρόβλημα. Σήμερα οι συμπολίτε στρέφουν το βλέμμα του μακριά από την Ευρώπη. Γυρίζουν την πλάτη τους στην Ευρώπη εξαιτία τη πολιτική που οδήγησε σε αυτές τις οδυνηρές ε, συνέπειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του εμπειρογνώμονε και να του ρωτήσω το εξή. Δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα, ευελιξία. Αναζήτηση βέβαια δημοσιονομικής ισορροπίας χρειαζόμαστε, αλλά τόση πολύ ελαστικότητα θα μπορούσαμε παράλληλα να εφαρμόσουμε και έναν κανόνα που θα λέει ότι όλοι οι, κανό, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ένα εισόδημα που θα είναι πάνω από το κατόφλι της φτώχειας. Να το εξασφαλίσουμε αυτό με έναν κανόνα γιατί έχουμε ακόμη και στη Γαλλία κανόνες που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχουμε δηλαδή πολιτικές που υποτίθεται ότι θέλουν να, να βοηθήσουν τον κόσμο να ε, ξεφύγουν από μια επισφαλή οικονομική κατάσταση, αλλά δυστυχώς δεν το καταφέρνουμε. Ο κύριος Σέρκας για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να θέσω μια ερώτηση σε κάθε έναν από τους παρεμβαίνοντες. Λυπούμε που έφυγε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γιατί, ξέρετε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έναντι αυτής της κατάστασης. Και δεν είναι έτσι. Έχουμε το άρθρο 154 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα του Συμβουλίου τη Ευρώπη, παρόλο που δεν είναι η ίδια συμβαλόμενο μέρο. Θα ήθελα να πω σε όλου ότι με εντυπωσίασε η άποψή του η άποψη όλων σας με εντυπωσίασε, ήταν πολύ πλουραλιστική. Δεν είναι το θέμα ε, ο διαχωρισμός μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αυτό το οποίο υπερασπιζόμαστε είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το μέλλον της Ευρώπης, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο εάν θα πρέπει οι άνθρωποι να υπηρετούν την οικονομία ή η οικονομία να υπηρετεί τις ανθρώπους, τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το διακύβευμα, είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όλοι οι παρεμβαίνοντες το ανέλησαν. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Πενέδα. Ως προς, ως προς τα προγράμματα αυτά, εγώ νομίζω ότι επιβλήθηκαν οι χώρες έχασαν ε, ε κυριαρχία, δεν μπορούσαν να ε, έχουν το δικό τους νόμισμα, προσχώρησαν στο κοινό νόμισμα και στη συνέχεια υπέπεσαν στον εκβιασμό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Πορτογαλία προσέφηκε στο Πορτογαλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο είδε ότι οι επιταγές της Τρόικας ήταν αντίκυντο, αν θέλετε, σε ε, συνταγματικές διατάξεις ε, της χώρας αυτής. Ως προς τον κύριο Ρέιμον Τόρες, θα ήθελα να του πω το εξή. Θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερο στο μέλλον όχι μόνο να κάνετε ανάλυση της κατάστασης, αλλά να παρουσιάζετε και εναλλακτικέ λύσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Κανείς δεν αρνείται εδώ τις μεταρρυθμίσεις και τη λιτότητα, αλλά να είναι χρήσιμες μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές, χρήσιμη λιτότητα η οποία ε, να γίνει για να λυθούν προβλήματα, όχι να δημιουργηθούν επιπρόσθετα. Ερωτώ λοιπόν, σας ε, ζήτησε ποτέ τη γνώμη σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο, εσείς που είστε εμπειρογνώμονες και έχετε συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα. Σας ζήτησαν ποτέ τη γνώμη σας, ε, σας κάλεσαν ποτέ να βοηθήσετε. Αυτό θέλω να μάθω. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι διαθέσιμη, διατίθεται να μας συνοδεύσει σε αυτό το εγχείρημα, να δώσουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή απάντηση ε, σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ενσωματώνοντας όλες τις προοπτικές και όλες τις πολιτικές, όχι μόνο τις οικονομικό ε, δημοσιονομικές αλλά και τις κοινωνικές και εργασιακές. Είστε, διατίθεστε, προτίθεστε να μας συνοδεύσετε έτσι ώστε ε, οι προσαρμογές, οι μελλοντικέ να λάβουν υπόψη τους και το κοινωνικό και εργασιακό σκέλος εσείς στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Και τέλος θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να κάνω το εξής σχόλιο. Έρχονται στιγμές στη δράση ε, των κοινοβουλίων που ε, είναι κρίσιμες και θα πρέπει να αντλήσουμε το δίδαγμα της Ευρώπης δεν αγιάζει ο σκοπός τα μέσα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε στον εκάστοτε σκοπό και νομίζω ε, ότι ε, δεν μπορεί κανείς ε, επειδή είναι αισιόδοξο ή βολονταριστής αν θέλετε να εφαρμόσει όποιο μέσο θέλει για να πετύχει το σκοπό του. Το μέσο πρέπει να είναι αναλογικό, έξυπνο, δημοκρατικό, όχι επιβλησέν. Αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες ε, ε, ενός πράγματος το οποίο είναι φρικτό, ε, ένα, μια νέα μορφή απολυταρχισμού, την οποία αντιλαμβάνονται υποτίθεται μόνο οι τεχνοκράτες και οι οικονομολόγοι. Νομίζω λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να ανακτήσει τη δημοκρατική του νομοποίηση και ευχαριστώ όλους όσοι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν όλα τα μέλη ε, που ήθελα να πάρουν το λόγο. Δυστυχώς ο κύριος Πέτρος Στάγκος δεν είναι πλέον στην αίθουσα, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους τρεις εμπειρογνώμονες που είναι παρόντες. Πρώτον, Χωσέ Σίλβα Πενέδα. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά δυστυχώς. Ε, Μόνο σας ζητώ να μην τα ξεπεράσετε αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθώ να είμαι λακωνικός και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Ρεζίνα Μπάστος, θα ήθελα να πω ότι παρά την κατάσταση αυτή, εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ικανότητα των Πορτογάλων και ιδιαίτερα των Πορτογάλων επιχειρηματιών ήταν αξιοθαύμαστη και αξιοσημείωτη. Και παρά τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης, ε, ε, επιβίωσαν πολλές οι επιχειρήσεις ε, και αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Ε, οι εξαγωγές της, Ιταλίας, της ε, Πορτογαλίας αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές της ε, Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας. Και παρόλο που το κόστος ενέργειας είναι πολύ υψηλό, Έχουμε δυνατότητε λοιπόν και υπάρχουν πολλέ θετικέ ενδείξει ότι θα ξεφύγουμε από την κατάσταση. Βέβαια ήταν τόσο σοβαρή η κρίση που σε καμία περίπτωση δεν θα ξαναεπιστρέψουμε ποτέ στο σημείο τη αφετηρία. Είναι λάθο πιστεύω ότι κάποτε θα γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση. Συμφωνώ ότι βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Και αυτή η ενδιάμεση φάση ε, χαρακτηρίζεται από πολλές ανισορροπίες και πολλές αδικίες. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση. Για να φτάσουμε στην επόμενη φάση θα πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος. Και το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέο δεν μπορεί να είναι ο μοναδικό στόχο, ούτε καν στόχο πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι μέσο. Ο βασικό στόχο είναι η μείωση τη ανεργία. Και θα πρέπει το ποσοστό ανεργία να είναι το πολύ 2%. Και τώρα πώς επιτύχουμε χαμηλό ποσοστό ενεργείας θα πρέπει να το δούμε με κοινωνικά μέτρα. Ε, η Νέζουμπερ ε, μίλησε για, για τη διάγνωση και τα λάθη. Έχει και ένα άλλο ελάττωμα το πρόγραμμα. Προσπάθησε να δημιουργήσει, να λύσει ταυτόχρονα δύο αντιφατικά θέματα. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να προσπαθεί να διορθώσει και το δημοσιονομικό έλλειμμα και την εξωτερική ανισορροπία. Είναι αδύνατο. Αυτή ήταν η παράδοση της Τρόικα ε, και δεν μπόρεσε να υποτιμηθεί νόμισμα γιατί δεν είχαμε δικό μας νόμισμα οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε άλλες μεθοδολογίες για να επιδιώξουμε τον ίδιο στόχο αλλά προσπάθησε να μειώσει το εξωτερικό έλλειμμα με τη μείωση των εξαγωγών. Τι έγινε όμως με την μείωση του εσωτερικού με τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης δεν μπορέσαμε ποτέ να καλύψουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Είναι αντιφατική λοιπόν αυτή η στόχη να επιδιώκονται ταυτόχρονα έχουμε μία άρρωστη κοινωνία. Ο γιατρός που ήταν η Τρόικα έπρεπε να κάνει τη διάγνωση της αρρώστιας και να βρει το σωστό φάρμακο. Εδώ ε, επιβλήθηκε ένα φάρμακο χωρίς να έχει γίνει η σωστή διάγνωση. Οπότε, παρόλο που κάποιες επιχειρήσεις και οι συνδικάτα πρότειναν κάποιες αλλαγές, Τρόικα έμεινε αδιάλακτη, αμετάβλητη και ανέστητη απέναντι στις εκκλήσεις των κοινωνικών εταίρων. Και αυτό πραγματικά είναι μια μαρτυρία που κάνω έχοντας γνώση της κατάστασης. Η Άννα Γκόμες μίλησε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν είμαι πια ευρωβουλευτής για να δώσω τέτοια απάντηση. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας. Ε, και για να απαντήσω στο σχόλιο του Τόμας Μάν, το θέμα της ουσίας είναι ότι είναι δυνατόν να έχουμε νέο νόμισμα σε μια ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζει σημαντικές ε, διαδροθετικές ανισορροπίες, έχει διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές κοσμοθεωρίες και όραμα για τον κόσμο. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή την ευρύτερη περιοχή ως τάμπουλα ράζα που όλα είναι ίδια και ομοιόμορφα. Οπότε να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα οικονομικής πολιτικής στο Νότο, στην Πορτογαλία και στο Βορρά είναι α, αντιφατικό και αντιβαίνει στο ίδιο το ευρωπαϊκό πνεύμα. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο για όλους, να κάνουμε αντιγραφή και επικόλυση του ίδιου μοντέλου σε όλους, γιατί οι συνέπειες, ιδιαίτερα οι κοινωνικές, είναι πολύ αρνητικές. Και παρά τις κριτικές που έγιναν, τίποτα δεν άλλαξε ε, στην ε, πορτογαλική οικονομία. Τώρα, τι θα σημάνει το τέρμα της Τρόικας. Ε, θα φύγει η Τρόικα και θα σταματήσει η λιτότητα. Όχι. Η αποχώρηση της Τρόικας ε, δεν θα σημάνει το τέλος της λιτότητας. Γιατί εξακολουθούμε να υποχρεώμαστε να συγκρατήσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα και να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Άρα θα χρειαστεί να, προσπαθεί, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε μέτρα και πάλι δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά θέλουμε να, να πετύχουμε μια οικονομική ανάπτυξη για να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Και έπρεπε και εμείς να έχουμε σημαντικό βάρος στη συζήτηση, ε, στη συζήτηση για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλιώς, αν δεν άβουμε εμείς μέρος στη συζήτηση και αν δεν είναι να παίξουμε ενεργό ρόλο στην λήψη της απόφασης, την απόφαση αντί για μας θα τη λάβουν οι γραφειοκράτες, οι τεχνοκράτες της Ευρώπης. Γιατί ταυτόχρονα έπρεπε να έχουμε τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική ανάπτυξη και ένα πολύ ευρύτερο ορίζοντα δεκαετή και όχι τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και ταυτόχρονα σε αυτή τη δεκαετία να επιδιώξουμε και την εξυγίανση την δημοσιονομική και των δημόσιων λογαριασμών. Αυτά ευχαριστώ. Λυπούμε, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Το λόγο έχει ο Ρεμόν Τόρε. Ευχαριστώ καταρχήν για την ε, εξαιρετική ποιότητα της συζήτησης και τα σημαντικά θέματα. Υπάρχει ένα σύνολο ερωτήσεων που άπτεται του λόγου συνέχισης των προσπαθειών αυτών, αφού τα αποτελέσματα είναι αυτά που είπαμε. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποια στοιχεία για μια απάντηση. Πρώτον, κάποιοι θεσμοί, ε, κάποιοι κανόνες ε, ε, του εργασιακού δικαίου εμπόδιζαν την ανάπτυξη. Υπήρχε μια γενική πρόσληψη κοινή προς αυτό, με αυτό το περιεχόμενο. Ε, και για, πιστεύω ότι τα άτομα τα οποία κλήθησαν να εφαρμόσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις προσαρμογές, δεν είχαν ε, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και γνώσεις. Ε, υπάρχει μια άλλη πρόσληψη. Το ότι δεν μπορούμε να επιφέρουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή παρά μόνο με τον τρόπο που αποφασίστηκε. Ε, δεν θεωρήθηκε δυνατό ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας διαφορετικός ρυθμός προσαρμογής και ένα διαφορετικό περιεχόμενο που θα ευνοούσε περισσότερο την απασχόληση. Το λέγαμε από το 2010, όχι από το 2009. Είναι ενδιαφέρον. Ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ένα τμήμα ερευνών ε, και με μία έρευνα που έγινε αναγνωρίστηκε ότι οι πολιτικές οικονομικής εξυγίανσης θα είχαν πολύ πιο αρνητικές συνέπειες για τις θέσεις εργασίας και για την ε, ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας δεν ελήφθησαν υπόψη, μόνο εκ των υστέρων αναγνωρίστηκαν. Άλλο στοιχείο, η οικοδόμηση του ευρώ μία ενιαία νομισματική ζώνη ε, απαιτεί και αντίστοιχους ενιαίους θεσμούς, μια ενιαία οικονομική και κοινωνική πολιτική. Οικονομική όσο αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα που μόλις φέτος αποφασίστηκαν και μια ε, ε, κοινωνική πολιτική. Μια νομισματική πολιτική δεν μπορεί παρά να βασίζεται και σε έναν κοινωνικό πυλώνα. Ένα άλλο, μια άλλη ερώτηση είχε να κάνει με το πώς να φέρουμε τον πληθυσμό ε, πιο κοντά, πώς να πείσουμε την κοινή γνώμη. Υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία εδώ. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουμε, ε, σε πολλές χώρες της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας η... δεν υπάρχει ισορροπία στις μεταρρυθμίσεις ε, και η κοινή γνώμη δεν αντιλαμβάνεται ε, όταν γίνονται πολύ απότομα οι μεταρρυθμίσεις και με ε, ευνίδιο τρόπο η κοινή γνώμη είναι αδύναμη να αντιληφθεί την αναγκαιότητά τους. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση όταν μια μεταρρύθμιση έχει όλο το χρόνο για να εφαρμοστεί. Δεύτερο στοιχείο. Η κοινή γνώμη χρειάζεται επίσης και το μακροπρόθεσμο όραμα. Φυσικά τα μέτρα αυτά, όπως είπε και ο κύριος Πενέντα, ελήφθησαν ε, ε, με βιασύνη, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι σήμερα διανύουμε ένα καινούριο στάδιο, όπου η μακροπρόθεσμη προοπτική λαμβάνει όλη τη σημασία που της αξίζει και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μακροπρόθεσμα προγράμματα για την οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία. Τρίτον, οι πληθυσμοί επίσης επιθυμούν συγκεκριμένες λύσεις στον τομέα χρηματοπιστωτικό ή τον οικονομικό τομέα υπήρξαν συγκεκριμένες ε, παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα τα ταμεία εγγυήσεων για την ανεργία των νέων. Αυτό δεν έγινε στον κοινωνικό τομέα. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για όλα τα νοικοκυριά ε, όπου είναι όλοι άνεργοι, και όπου υπάρχει μια συνιστός φτώχεια πάρα πολύ ανησυχητική μια, άλλη ερώτηση, νομίζω του Αλεχάντρο Θέρκας, ε, αφορούσε τους τυχόν αναλλακτικού τρόπους ε, και κατά πόσο υπήρξε διαβούλευση. Ε, νομίζω απαιτείται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νομίζω ότι αυτό υπήρξε στο παρελθόν και ότι εδραιώθηκε περισσότερο ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης, μόνο που σε σχέση με τα μέτρα που έλαβε η Τρόικα, οφείλω να ομολογήσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δεν συμμετείχε, δεν ε, τη συμβουλεύτηκαν ε, η Τρόικα όταν, κατα... Ε, καταστρώνει αυτά τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής ε, θα πρέπει ίσως να δέχεται και μια δεύτερη άποψη, μια εναλλακτική πρόταση ή να υπάρχει ένας περιοδικός μηχανισμός παρακολούθησης, καταγραφής των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης, ίσως κάθε έξι μήνες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο τελευταίος εμπειρογνώμονας, ο κύριος Τόρσεν, έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις αλλά και τη συμβολή σας στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω. Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα όσον αφορά στην Τρόικα. Η δημοκρατική, της νομιμοποίηση, οι κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις και το κατά πόσο αυτά τα μέτρα έχουν οικονομικό νόημα. Αυτά τα τρία μας ενδιαφέρουν. Από πλευράς δημοκρατικής νομιμοποίησης νομίζω ότι είναι σαφέστατο και στηρίζω το κείμενο που έχετε συντάξει ότι μέσα στη δομή της Τρόικας Σίγουρα υπάρχουν υποδομές που έχουν μειώσει το δημοκρατικό έλεγχο, τον έχουν περιορίσει και άρα ε, γύρεται το ερώτημα τι ε, σημαίνουν όλα αυτά για θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία δεν έχει καμία εντολή να παρέμβει στην αγορά εργασίας ωστόσο με τις αποφάσεις της την επηρεάζει άμεσα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ε, απεικονίζεται και πώς απεικονίζεται αυτό στην έκθεση και θα πρέπει αυτό το θέμα πολιτικής να το δουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο απαιτεί την υψηλή συνεισφορά, μεγάλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η σωστή άγουσα. Και άλλωστε η συνέπειε ήταν καταστροφικές σε κοινωνικό και εργασιακό πεδίο. Αυτό είναι σαφέστατο, νομίζω ότι το παρατηρούν όλοι και ως εκ τούτου η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι ε, υπάρχει και εξασφαλίζεται όταν ε, αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και τα επιλύνουμε αποτελεσματικά. Σίγουρα οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό πρέπει να το λύσουμε με τις ε, ομιλίες και τις εκφωνήσεις ομιλιών δεν πρόκειται να το επιλύσουμε πρέπει να αναλυφθεί δράση. Το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με το κατά πόσο τα μέτρα αυτά έχουν οικονομικό νόημα. Δουλεύουν, ναι ή όχι, είναι λειτουργικά, ναι ή όχι. Νομίζω ότι οι ομιλητέ συμφωνούν. Οι μεταρρυθμίσει δεν είχαν οικονομικό αντίκτυπο, δεν είχαν οικονομικό αποτέλεσμα. Ω προ τι μισθολογικέ περικοπέ, φάνηκε ξεκάθαρα ότι όσο περισσότερο μειώνονται οι μισθοί, θεωρείται ότι οι επιχειρήσει θα γίνουν πιο ανταγωνιστικέ, θα εξάγουν περισσότερο και θα υπάρξει ένα σωρό ανάπτυξη. Όμω, περικόπηκαν οι μισθοί και μάλιστα πολύ, χωρί να υπάρχει αύξηση των θέσεων απασχόληση, ούτε αύξηση των εξαγωγών και τη ανταγωνιστικότητα. Οι μελέτε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι αυτή η σχέση ε, σύμφωνα με την οποία μειώνονται υποτίθεται οι τιμέ γιατί έχουν μειωθεί οι μισθοί και άρα θα μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη εξαγωγή των προϊόντων κτλ. Οι ίδιε οι μελέτε του ΔΝΤ δείχνουν ότι αυτό δεν λειτουργεί. Το μόνο που κάνει είναι οι επιχειρήσει να βελτιώνουν το περιθώριο κέρδου του και τίποτα άλλο. Λάθο είναι το σημείο στο οποίο έχουμε στρέψει, έχουμε εστιάσει την προσοχή μα Να μην συγχαίουμε αυτά τα δύο σε όλες αυτές τις χώρες. Και επαναλαμβάνω το κάλεσμά μου, την έκκληση που απευθύνω. Έχουμε θεσμούς και όργανα συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες μέλη. Οι ε, ε, θεσμούς συλλογικότητε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις που έχουν υποστεί τεράστιες πιέσεις από την Τρόικα έχουν μειωθεί τα μέλη τους. Κατά, ε, το 1 τρίτο, για παράδειγμα, έχει μείνει στην Πορτογαλία. Σαφέστατα πλέον το να εστιάζει κανείς την προσοχή του μόνο στην ανταγωνιστικότητα και στο να ασκεί πίεση να περικοπεί και να περιοριστεί το μισθολογικό κόστος είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί. Ε, και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ήταν υποδειγματική στη δουλειά της μέχρι σήμερα. Υπάρχει άλλο μοντέλο που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική ισότητα και πρέπει να αξιοποιηθεί και να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Και σας δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα πριν τελειώσει ο χρόνος μου. Έχουμε δει για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία λοιπόν θέσπισε ένα σύστημα το οποίο συζητείται σήμερα και στη Γερμανία βλέπουμε τις ε, διαπραγματεύσεις στη Γερμανία, στις συλλογικέ, στις εργασιακές που πηγαίνουν προς μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση πλέον σε σχέση με το παρελθόν. Η Γερμανία είδε ότι πάρα πολύ λίγες συλλογικές συμβάσεις είναι δεσμευτικές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία με καλύτερο τρόπο. Και άρα η γερμανική κυβέρνηση ασκεί πίεση για την έλευση μεταρρυθμίσεων μέσα στην, ε, ίδια τη Γερμανία, μέσα στη χώρα αυτή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ απεριόριστα και τους τέσσερις καλεσμένους μας για τη δημόσια αυτή ακρόση που ήταν ε, συναρπαστική, μερικές φορές απογοητευτική για μερικές δηλώσεις, αλλά σίγουρα πολύ επικοδομητική για την αξιολόγηση του έργου της Τρόικα, για τον αδιέξοδο που οδήγησε μερικές μεταρρυθμίσεις ε, στο κοινωνικό τομέα. Και δυστυχώς ε, μας οδείξαν και στην πεποίθηση ότι το άρθρο 9 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Είμαι βεβαία πάντως ότι υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση του εισηγητή μας του κυρίου Σέρκας θα ληφθούν, θα ληφθούν δεόντως υπόψη οι παρατηρήσεις για τις οποίες σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώσαμε αυτή τη δημόσια κρόση. Μας έχουν απομείνει όμως δύο καλεσμένοι, από τους οποίους ζητώ ειλικρινά Συγγνώμη για την ε, αρκετή καθυστέρηση που είχαμε πάνω από μισή ώρα και παρακαλώ τους συναδέλφους που φεύγουν από την αίθουσα να αποχωρήσουν ήσυχα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Φρεντερίκ Νταρντέν που τηλεγραφικά θα μας ενημερώσει για τις χθεσινές διαπραγματεύσεις ε, με την Ελληνική Προεδρία ε, για το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας, της ενίσχυσης συνεργασίας ε, μεταξύ των ε, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Κύριε Νταρντέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χθε είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο με αυτό το θέμα και παρά από πεντά ώρες διαπραγματεύσεις ε, δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε κανένα συμπέρασμα δεν είχαμε σημαντικές πρόοδους, αλλά μην είμαστε απεσιόδοξοι. Μερικές διευκρινήσεις. Καταρχήν, εκούσιος ή υποχρεωτικός χαρακτήρας της συμμετοχής των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στο δίκτυο. Η εντολή της, της Επιτροπής μας ήταν σαφής και κατηγορηματική. Εμείς ταχθήκαμε υπέρ της θέσης για υποχρεωτικό χαρακτήρα της συμμετοχής στο δίκτυο. Αυτή ήταν η δική μας εντολή, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο για περισσότερο πολιτικούς παράνομικούς λόγους ε, έχει διαφορετική θέση. Από την ανταλλαγή απόψε διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν βάσιμα νομικά κολλήματα, περισσότερο ήταν πολιτική η θέση. Θα δούμε τι πρόοδο θα δημιουργηθεί στο... στη συνέχεια. Τώρα, η παρουσία του Συμβουλίου στο δίκτυο ΕΜΚΟ ε, στη θέση του παρατηρητή. Εμείς ε, θελήσαμε ε, να συμφωνήσουμε για την παρουσία αυτή με την ιδιότητα του ε, παρατηρητή, υπό τον όρο όμως της υποχρεωτικής συμμετοχής στο δίκτυο και ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λειτουργία του δικτύου, το Συμβούλιο θέλει να προσδιορίσει τους όρους της άσκησης και της ανταλλαγής στη βασική πράξη και τα υπόλοιπα να τα αφήσει στις αρμοδιότητες του δικτύου. Εμείς υποβάλαμε μια εναλλακτική πρόταση και μάλιστα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαμε ότι θέλουμε στη βασική πράξη να διατηρηθούν κάποια θέματα όπως προσαρμογή με βάση τους στόχους που επαναδιαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο, όλα αυτά στη βασική πράξη, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε κατά εξουσιοδότηση πράξη για να μπορέσουμε, χάρη ευελισία και ελαστικότητα, να προσαρμοστούμε στι νέε εξέλιξει. Σε ό,τι αφορά την αποστολή του δικτύου, καλή ιδέα, αλλά κάποια στοιχεία όπως οι δείκτες και η μεθοδολογία του bench learning θα πρέπει να παραπευθούν στις κατεξουσιοδότηση πράξεις, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτά τα τρία σημεία η Ελληνική Προεδρία θα μεταφέρει τη θέση μας στο, στην Κορεπέρ για να δούμε το περιθώριο λιμών του Συμβουλίου. Τώρα, το θέμα του ορισμού του bench learning είναι σημαντικό. Θέλουμε επίσης μια σαφή συμμετοχή που θα είναι εθνική και αυτόματη των δημοσίων ε, υπηρεσιών απασχόληση στο δίκτυο. Επίση αναφέρεται η εθελούσια κινητικότητα, η εφαρμογή τη στρατηγική του 2020, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η καταπολέμηση της ανεργία, ε, η λήψη υπόψη των πιο ευάλωτων ε, ανέργων όπω των νέων των ηλικιωμένων. Για τα σημεία αυτά είχαμε σημαντικέ προόδου. Και τέλο, ό,τι αφορά τη νομική βάση, η αναφορά του άρθρου 14 Εκεί προτείναμε μια νέα διατύπωση μετά από τις νομικές γνωμοδοτήσεις και η διατύπωση αυτή θα σας μοιραστεί στο μέλλον, στις επόμενες μέρες, ώστε να μπορέσει η Ελληνική Προεδρία να παρουσιάσει στην Κορεπέρ της 17ης του μηνός όλα τα στοιχεία και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευελπιστούμε στις 22 του μηνός θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για αισθητές ε, εξέλιξεις και πρόοδο, ώστε να ολοκληρώσουμε 22-29 και να διαθετηθεί το θέμα στην Ολομέλεια του Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της καταπολέμησης ανεργίας ε, ε, Ελπίζω ότι και χάρη σε κάποιες άλλες συμφωνίες θα καταλήξουμε τελικά σε αίσιο πέρα. Σας Ευχαριστώ για την πιστή αυτή παρουσίαση του χθεσινού τριμέρους διαλόγου. Ήταν πραγματικά εκτενέστατη και πολύ περιστατωμένη παρουσίαση. Εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω και δεν έχουμε και ερωτήσεις για το θέμα αυτό, οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο της ενημέρωσης για το τριμερή διάλογο και ζητώ και πάλι συγγνώμη από τους καλεσμένους μας γιατί καθυστερήσαμε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων του σημείου 6. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με τον Ντομά Ντομινίκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, και τον Τόμ Μπέβερς, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, της ΕΜΚΟ δηλαδή, και SPC είστε πολύ σημαντικοί φορείς και οι δύο και οι δύο επιτροπές στα πλαίσια της δικυβέρνησης της Ευρωζώνης, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού πυλώνα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, μέχρι στιγμής είχαμε λίγες επαφές και γι' αυτό θέλησαμε να οργανώσουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση. πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, το Ευρωπαϊκό Εξαμήνιο και το θέμα τη ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Λυπούμε όμω γιατί αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, αλλά έχουμε εκπροσώπου ε, από όλε τι πολιτικέ ομάδε και θα μεταφέρουν ε, και στου συναδέλφου του αυτά που θα ακούσουν εδώ. Θα δώσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο στον καθένα Δυστυχώς ε, οι ευρωβουλευτές δεν είναι εξοικειωμένοι με τους φορείς, με τις δύο επιτροπές ε, που εκπροσωπείτε. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσετε για τη συμβολή των δικών σας ε, επιτροπών σε αυτόν τον κύκλο και να μας δώσετε κάποιε προοπτικές για το έργο σας. Ακούσατε από τον Φρεντερικ Νταρντέν την ενημέρωση από τον χθεσινό τριμερή διάλογο για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο θέλει να συμπεριλάβει το ΕΜΚΟ στην δομή αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που ίσως έχουμε την ευκαιρία, ίσως έχουμε την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε, έχει κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη συμπερίληψη αυτή. Αυτά λοιπόν, θα δώσω πρώτο λόγο στον Τωμά Ντομινίκ και να τα καθακούσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας παρόλο που είναι διαφορετικέ οι λειτουργίε των δύο επιτροπών. Ο Στομάτο Μινίκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και που διοργανώσατε και αυτήν τη συνάντηση. Ε, θα προσπαθήσω να μιλήσω διαρθρωμένα πάνω στο θέμα που μας αφορά, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το συντονισμό των πολιτικών. Επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές να παρουσιάσω την Επιτροπή μου. Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, SPC. Η κύρια αποστολή της είναι να εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο στα θέματα της κοινωνικής προστασίας, να παρέχει συμβουλευτικές γνώμες. Θα ξεκινήσω με την κοινωνική διάσταση. Η κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, ε, που είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον πολίτη. Το είδαμε και στη σημερινή συζήτηση. οι περισσότεροι κοινωνικοί δείκτες έχουν χτυπήσει κόκκινο, κανέναν δεν θα καταπλήξει αυτό. Όπως λέει η Ευρωστάτ, τα επίπεδα της φτώχειας ε, το 2012 ήταν τα υψηλότερα ποτέ, πολύ άσχημοι δείκτες φτώχειας ε, και κοινωνικού αποκλεισμού. Από το 2010 σταθερά αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών. σε μερικές χώρες υπερβαίνει το 2% ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, ε, οι, συνθήκες, οι οικογένειες που τελούν σε συνθήκες ε, επισφάλειας επιδεινώνονται. Όλες αυτές οι τάσεις επιβεβαιώνονται από τους δείκτες επιδόσεων κοινωνικής προστασίας. Ε, το καθεστώς τους είναι καθεστώς παρακολούθησης. Αυτόν τον όρο χρησιμοποιούμε. Προσπαθούμε να έχουμε συζητήσεις και δείκτες για τις κοινωνικές πτυχές και για την επίπτωση κάποιων μεταρρυθμίσεων και βάσει αυτών να επεξεργαστούμε δείκτες. Ε, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε όλα εκείνα, όλους εκείνους τους τομείς που έχει να κάνει με τις συνθήκες της φτώχειας, της οικογένειας, τα νοικοκυριά, τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος της μισθολογικής πολιτικής για να ανατρέψουμε τις υφιστάμενες τάσεις. Αλλά ο κύριος όρος για την ανατροπή των περιστάσεων αυτών είναι οι κοινωνικές επενδύσεις και η ανάπτυξη. Και πρόσφατα έχουμε το λεγόμενο scoreboard, πίνακα επιδόσεων, το οποίο είναι ένα εργαλείο που υιοθετήθηκε τον περασμένο χρόνο η Επιτροπή μου συνέστησε στο Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιμένοντας όμως ότι η επιλογή των δίκτων θα πρέπει να οδηγήσει σε αναθεώρηση των όσων έχουμε εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Μας ενδιαφέρει επίσης ο συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, δεδομένης και της έντασης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αντιπροσωπεύουν το 29% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, του ΑΕΠ της Ένωσης. Απέναντι στην ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, λόγω και της κρίσης, υπάρχει μία μέθοδος που ονομάζεται MOC στα γαλλικά, OMC στα αγγλικά, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Είναι η ομόνη μορφή συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών σε επίπεδο ένωσης. Και αυτό σε ένα πλαίσιο όπου αυξάνονται οι εθνικές αποκλήσεις. Όπως το ξέρετε η μέθοδος αυτή είναι μια μορφή συντονισμού που βασίζεται στην ε, δέσμευση των κρατών μελών. Είναι θελοντική. Θέλω να προσδιορίσω ότι να, να διευκρινίσω μάλλον, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει καταστήσει δυνατή τη λήψη πρωτοβουλειών για τον συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών δεν σημαίνει εναρμόνιση της κοινωνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Αυτό απαγορεύεται νομικά στην Ένωση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, απομένουν ελεύθερα ε, να βρουν εκείνα τον, τον επιθυμητό συμβιβασμό μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης. Τέλος, κάποιες παρατηρήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Από το 2011 συμμετέχουμε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης στην προετοιμασία της απόφασης του Συμβουλίου και στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Παρατηρούμε ότι σιγά σιγά γινόμαστε ένα κέντρο δημόσιου συντονισμού, συντονισμού των δημόσιων πολιτικών, όπου υπησέρχεται επίσης η υγεία και η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις στατιστικά στοιχεία, 28% των συστάσεων που υιοθετήθηκαν το 2013 αφορούσαν την κοινωνική προστασία, τη σύνταξη, την υγεία, την ε, καταπολέμηση της φτώχειας, ε, την λειτουργία της κοινωνικής προστασίας. Αυτές οι δημόσιες πολιτικές ε, συντονίζονται λόγω της δημοσιονομικής πτυχής που έχουν μέσω των νομικών βάσεων που δεν δημιουργήθηκαν όμως για αυτές τις πολιτικές, άρθρα 121 και 148. Υπάρχει όμως μία αμφισβήτηση στις κοινωνίες. Το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί και θα το συζητήσουμε και αύριο. Η υλοποίηση των ε, μέτρων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων. Εμείς θέλουμε οι πολιτικές αυτές να συζητούνται από τους αρμόδιους υπουργούς στα αρμόδια συμβούλια. Δεδομένου του, τη δεδομένη σημασίας του ρόλου του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ με τους ε, τρεις κλάδους του στην ε, διαδικασία υιοθέτηση ε, των, των συστάσεων, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια πραγματική πλέον εστίαση στον πληθυσμό. Ε, υπάρχει πλέον ε, μια πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά ζητήματα όπως ακριβώς έχουν αντιμετωπιστεί τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Τόμ για την ΕΜΚΟ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από το 1998 η Επιτροπή Απασχόλησης που έχει παρόμοια σύνθεση με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας είναι το βασικό όργανο που προετοιμάζει το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, βάσει του σχετικού άρθρου της συνθήκης. Αυτή τη στρατηγική την έχουμε κατοχυρώσει με τη στρατηγική της Λισαβόνας στην Ευρώπη για το 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. 15 χρόνια λοιπόν έχουμε εμπειρία στο συντονισμό πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών ώστε να συγκλίνουν και να είναι αποτελεσματικές. Άλλωστε σήμερα δεν ταιριάζει το ίδιο κουστούμι σε όλους. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Προετοιμάζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, βασικά μηνύματα των εκθέσεών μας ε, συντάσσουμε. Ε, αναθεωρούμε τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα των κρατών μελών και άπαξ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει τις συστάσεις αναχώρα, τι συζητούμε και όταν χρειάζεται τις τροποποιούμε πριν ε, γίνουν ε, συστάσεις του Συμβουλίου του Ιουνίου. Έτσι δουλεύουμε λοιπόν. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς παρακολουθούμε την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα μέσω μιας διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας για να υπάρξει αντικειμενικότητα. Είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτήν. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και κάνουμε peer review, αναθεώρηση ομολόγων. Τις εξελίξεις ε, τις συζητούμε σε βάθος, με ευρύ πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, έλαβαν χώρα. Η διαδικασία μας πάντοτε βασίζεται σε στοιχεία που θα πρέπει να συγκεντρώσουμε για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα και πάντοτε συμπεριλαμβάνουμε αναφορά στην ε, απασχόληση των νέων. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο. Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με άλλους τομείς της αγοράς εργασίας και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα ασχοληθούμε και με τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας. Έχουμε σχέδιο συστάσεων που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική μας Επιτροπή και ε, όλες αυτές τις θέσεις και τις αλλαγές τις ενσωματώνει το Συμβούλιο. Από τότε που ξεκίνησε η στρατηγική για την Ευρώπη το 2020, η δική μας Επιτροπή είναι πεπισμένη για το ότι η δουλειά μας είναι αν όχι το ίδιο ποιοτική μπορεί και παραπάνω και περισσότερο ποιοτική από άλλους σχηματισμούς του Συμβουλίου και μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ και αυτό έχει συμβάλει στο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο καλύτερο και να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική δεν είναι παράπλευρη απώλεια ή παρενέργεια, θέλετε, των αποφάσεων που εφαρμόζονται στο οικονομικό πεδίο. Αντιθέτως, τα θέματα αυτά είναι στον πυρήνα του προς τα που θα πρέπει να πηγαίνει η Ευρώπη και θα πρέπει να ενισχύσει και το κοινωνικό σκέλος της ΟΝΕ. Είμαστε πεπισμένοι ότι τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να την κάνουμε με βάση την υφιστάμενη εμπειρία ε, σε θέματα ευρωπαϊκής απασχόλησης με τη συμβολή όλων των κρατών μελών ε, και φυσικά όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ. Έχουμε ε, πολυμερή εποπτεία και μπορούμε πάνω σε αυτή να χτίσουμε καλύτερο συντονισμό εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, προληπτικούς, κατασταλτικούς ελέγχους για να είμαστε αποτελεσματικοί και αν χρειάζεται περισσότερη δουλειά εκ των προτέρων μπορούμε ως Επιτροπή να την κάνουμε, εάν χρειάζεται εκ των υστέρων μπορούμε να συμβάλλουμε και σε αυτό τον έλεγχο. Όλα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πολυμερή προσέγγιση, διότι έτσι όλα τα κρατημέλη μπορούν το καθένα να βάλει το λιθαράκι του, να εκφράσει την άποψή του, να υπάρξει νομιμοποίηση και ιδιοκτησία, αν θέλετε, κυριαρχία. Δεν μπορεί ένα θεσμικό όργανο να αντικαταστήσει δεκαετίες εσωτερικής γνώσης και εμπειρίας σε 28 κρατημέλη. Πράγματι, η Τρόικα στερεί το εμπειρία σε θέματα ε, πολιτικής απασχόλησης και αυτό είναι ένα εύγλωτο παράδειγμα του επιχειρηματός μου. Συγκεκριμένο βήμα για την ενίσχυση του κοινωνικού σκέλους είναι το εξή. Συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή Πολιτι... Κοινωνικής Προστασίας για πρόταση απασχόλησης και βαθμολόγιο, scoreboard. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014. Είναι ένα καλό σημείο κίνησης, όχι άφηξης και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, ε, να δουλεύουμε έτσι ώστε να έχουμε κοινέ εκθέσεις με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Το scoreboard, το βαθμολόγιο, έχει ενσωματωθεί πλήρως στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. και λειτουργεί ως μηχανισμός πυροδότησης έτσι ώστε να υπάρξουν αυτόματα συστάσεις προς τα κράτη-μέλη αλλά και να μελετηθούν ε, ακόμα περισσότερο τα υπάρχοντα στοιχεία. Ο συνάδελφος ανέφερε την παρακολούθηση των επιδόσεων σε θέματα κοινωνικής προστασίας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Έχει αποδείξει την αξία του και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε έτσι περαιτέρω. Βελτιώνουμε τη συνεργασία μας και με τους κοινωνικούς εταίρους, διαβουλευόμαστε με αυτούς σε κέρια σημεία κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα τελευταία χρόνια η συζήτησή μας έχει γίνει πιο ανοιχτή, πιο εμπλουτισμένη, λιγότερο τοπική. Η κοινωνική λιγότερο τυπική, με συγχωρείτε, η κοινωνική εταίρη είναι πολύ σημαντική και χρειαζόμαστε εθνικά μεταρρυθμιστικά στη σχέδια μόνο εάν έχουν καταρτιστεί ως αποτέλεσμα διαλόγου και συνένεσης. Χρειαζόμαστε κοινωνικό διάλογο πιο αποτελεσματικό, ε, πιο ενιαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορούμε όλα αυτά να τα πετύχουμε εάν συνεργαστούμε με τους κοινωνικούς εταίρους και θα το πράξουμε βεβαίως. Η ΕΜΚΟ, η Επιτροπή αυτή, θέλει να βελτιώσει τη συνεργασία της με το δίκτυο ε, δημοσίων υπηρεσιών για την απασχόληση. Θα πρέπει το δίκτυο αυτό να λάβει μια πιο επίσημη μορφή. Αυτό θα διευκολύνει και τη δική μας δουλειά και γι' αυτό θέλουμε να συνδεθούμε στενά με, την, με εκείνους. Ε, θα πρέπει να επιτευχθεί το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ δικτύου και δικής μου επιτροπής, να είναι σαφέστατος ο, ο ρόλος του κάθε και θα πρέπει τα, ε, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία έτσι όπως αυτή μεταφέρεται από ε, το χώρο εργασίας, από την πραγματικότητα, από αυτό το οποίο γίνεται στην πράξη. Με όλα αυτά μαζί θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τον κανονισμό και ως, Επιτροπή βεβαίως συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους ε, ε συνήθεις συνεργάτες μας έχουμε προβλέψει την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020. Έχουμε ξεκινήσει ένα απολεγισμό. Θα παρουσιάσουμε έκθεση τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις διάφορες μεταρρυθμίσεις της φιλόδοξης που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω ότι θα μιλήσουμε και για την εμπειρία που έχουμε ήδη όλοι αποκτήσει ε, έτσι ώστε να μην επιστρέψουμε ποτέ στο παρελθόν όπου η προσέγγιση ήταν απολύτως διμερής μεταξύ κράτους μέλους και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Όλα αυτά θα τα δούμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για το 2020. Θα μπορούσα να είναι πιο φιλική προς το χρήστη. Ε, και να πούμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι ελάχιστες δεσμεύσεις που οφείλουν να τηρήσουν τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική, καλύτερες επιδόσεις, benchmarking, δείκτες, όλα αυτά είναι εργαλεία, έχουμε εμπειρία, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πλέον. Παρακολουθούμε ε, την υλοποίηση του προγράμματος της εγγύησης στους νέους, ε, του γνωστού αυτού προγράμματος και έτσι Άλλωστε σας είπα ότι στις αρχές του περασμένου ε, ε, Δεκεμβρίου είχαμε ειδική συνάντηση για την ανεργία των νέων με αυτό το αντικείμενο μόνο. Και αυτές οι 28 διαφορετικές εγγυήσεις για τους νέους θα είναι ένα ε, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Θα στείλουμε μήνυμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Λίγα λόγια λοιπόν για το άμεσο μέλλον. Ε, ξεκινά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014 με κάποια ίχνη ανάκαμψης. Η αγορά εργασίας όμως παραμένει εξαιρετικά ευπαθής, ασταθής, κάτι το οποίο ε, αποδυναμώνει τη ζήτηση, πλήττει την ανάπτυξη και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάθος χρόνου από τη στιγμή που πολλοί χάνουν δεξιότητες και δυσκολεύονται να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας όπου θα τις ξανααποκτήσουν και θα τις τελειοποιήσουν γίνονται ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συνεχιστούν, θα πρέπει να επιταχυνθούν ενδεχομένω σε ορισμένε περιπτώσει, ωστόσο η προσπάθεια χρειάζεται χρόνο για να φέρει καρπού και δεν θα βελτιωθεί κατά πάσα πιθανότητα βραχυπρόθεσμα η κατάσταση στην αγορά εργασία, ενώ θα είναι όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις οι επιθυμητές. Σας ευχαριστώ. Θερμά ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους μας. Πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις τους και ευθυγραμμίζονται και με το δικό μας έργο. Θα δώσω το λόγο σε όλους όσους τον ζήτησαν. Για Ζωβιέτσκα, Σέρκας και Πρόεδρος, κατά εξαίρεση. Αυτή. Η κυρία Γεζοβιέτσκα, η πρώτη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οι φορείς σα ε, κάνουν μελέτες, αναλύσεις, προετοιμάζετε συστάσεις και γνωμοδοτήσεις. Ερωτώ, τι λάθη γίνονται από τα κράτη-μέλη στην κοινωνική πολιτική, γιατί στην προηγούμενη δημόσια κρόαση ακούσαμε για κάποια λάθη. Θα ήθελα όμως και εσείς να μου πείτε τι λάθη γίνονται από τα κράτη-μέλη, τι λάθη έχετε εντοπίσει εσείς στις επιτροπές σας γιατί βλέπουμε ότι οι πολίτες γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Η μεγάλη ελαστικότητα στο τομέα εργασίας ε, δεν φέρνει αποτελέσματα και εφαρμόζεται περισσότερο, ερμηνεύεται από τον επιχειρηματία προς δικό του όφελος. Τι λάθη από αυτά που εντοπίσατε θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποκλείσει, τι λάθη μπορούμε να βελτιώσουμε και τι δραστηριότητες, τι μέτρα θα πρέπει να αναλάβουμε προκειμένου να αποτρέψουμε ή να διορθώσουμε τέτοια λάθη. Και σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση, ποιε είναι οι προσδοκίε σα από τι κοινωνικέ πολιτικέ των κρατών μελών, τι πρέπει να κάνουμε ώστε η κοινωνική διάσταση να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίση, για να το καταλάβουν και οι συμπολίτε μας. Και σε ό,τι αφορά και πάλι την κοινωνική διάσταση, θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο θα έπρεπε η πολιτική οι πολιτικοί θύνοντες ε, και όσοι εφαρμόζουν την πολιτική να επικοινωνήσουμε τον κόσμο ώστε όλες οι μεταρρυθμίσεις αυτές να γίνουν αντιληπτές από τους πολίτες να είναι διαφανείς ε, και στο μέτρο του δυνατού να γίνουν αποδεκτές αυτές οι μεταρρυθμίσεις από τους πολίτες. Γιατί η τέξη του τάγκο, όπως λέμε, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να χορέψουν τάγκο, Οπότε θα πρέπει να γίνονται τα βήματα και από τους δύο, ε, να συμπαραταχθούμε τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικότερα να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ, Αλεχάντρο Σέρκας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, είχαμε μια πολύ σκληρή συζήτηση και έχουμε με την δεύτερη αυτή ακρόαση μια συνέχιση τη ίδια κατάσταση και των ίδιων ανησυχιών και μια καταστροφική κατάσταση στην Ευρώπη, αν και σε μερικέ χώρε είναι πιο καταστροφική από ό,τι σε άλλε. Και οι χώρε που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα για λήψη αποφάσεων, ευτυχώ για αυτέ, βρίσκονται στην καλή πλευρά του νομίσματο, στην καλή όψη του νομίσματο. Και οι χώρε που έχουν τι λιγότερε δυνατότητε είναι αυτέ που αντιμετωπίζουν την δυσχερότερη κοινωνική κατάσταση. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις ε, προσπάθειές σας, ε, το έργο των επιτροπών σα και τις ομιλίε που μας κάνατε. Και έχω μια ερώτηση. Η συνθήκη λέει ότι είστε όργανα που παρέχουν ε, γραμματοτήσει και συμβουλές προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Παρέχετε συμβουλές λοιπόν... Ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συμβουλές σας ή μόνο ε, το Συμβούλιο από συγκεκριμένη μορφή του Συμβουλίου Υπουργών ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και μόνο ο Επίτροπος Άντορ που είναι αρμόδιος για κοινωνικά θέματα. Γιατί μόνο για τομεακά θέματα ζητούν τη γνωμοδότησή σας. Η βασική, η πρωταρχική μας πρόκληση είναι να σταματήσει η κοινωνική πολιτική να είναι η σταχτοπούτα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα πρέπει να φέρουμε την κοινωνική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάνετε πολλές προσπάθειες, ε, έχουμε μεγάλη πρόοδο και πιστεύω, όπως λένε και πολλοί, ότι Ακριβώ επειδή έχουμε μια Ευρώπη των 28, είναι πολύ πιο δύσκολο να λάβουμε αποφάσει και σε κοινωνικά θέματα, όπω γινόταν στη δεκαετία του 80. Υπάρχουν ε, αρκετά φρένα. Αλλά με τι νέε μορφέ οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση έχουμε πραγματική ευκαιρία να έχουμε πραγματική κοινωνική διάσταση τη οικονομική διακυβέρνηση. Και αν αναγάγουμε την ε, κοινωνική πολιτική και την απασχόληση οι βασικέ μα προτεραιότητε. Έχω όμω μια ερώτηση. Κάνουμε συστάσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τις προετοιμάζετε και εσείς. Οι συστάσεις όμως είναι σαν να ζητούμε ελλημοσύνη από τους φτωχού, δηλαδή ελάχιστα λαμβάνουμε. Γιατί είναι άνθρωποι που βρίσκονται με το νερό πάνω από τη μύτη του ουσιαστικά και ζητούμε επενδύσει ε, ε, και ζητούμε χρηματοοικονομικές ροές, ενώ οι, οι αποφάσεις για την τόνωση της οικονομίας βρίσκονται σε άλλα χέρια δηλαδή να ε, υποβάλουμε συστάσεις ε, στα κράτη που βρίσκονται στη δινή οικονομική κατάσταση χωρίς να τους δίνουμε μέσα για να υλοποιήσουν αυτές τις συστάσεις ε, μας οδηγεί αναπόφευκτα σε διέξοδο. Τώρα ετοιμάζουμε τις νέες συμβάσεις. Αν με αυτές υποβάλλονται νέοι όροι και προϋποθέσεις, μια κατάσταση που είναι ήδη δυσχερής θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί που πλήττονται από την έλλειψη πόρου να είναι αυτοί που θα πρέπει να βρουν και τις λύσεις. Η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού που είναι ακούσια θεωρείται ότι είναι σωστή ή μπορούμε να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο στο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη οικονομική διακυβέρνηση να δώσει τα κράτη-μέλη κάτι περισσότερο από απλέ συστάσει, να του δώσει και λύσει. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Για μια φορά έχω κι εγώ πολλές ερωτήσεις να θέσω και εποφελούμε της απουσίας άλλων συναδέλφων για να το κάνω. Πριν όμως, σύμφωνα με το θεσμικό μου ρόλο, να υπενθυμίσω στον κύριο Σέρκας ότι η ΠΕΣΚΕ και η ΙΜΚΟ είναι επιτροπές που προβλέπονται από τη συνθήκη, όπως ακριβώς και η ΕΚΟΦΗΝ για την Νομισματική, Οικονομική και Πολιτική Επιτροπή. και υπάρχει το άρθρο 150 της συνθήκης η Επιτροπή Απασχόλησης έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών. Το άρθρο 150 της Συνθήκης διευκρινίζει ε, όλη την αποστολή της Επιτροπής, ε, ε, ενώ οι αρμοδιότητες της Ένωσης προσδιορίζονται στο άρθρο 9 της Συνθήκης σε σχέση με τις πολιτικές απασχόλησης. Επιτροπή Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας, ε, παράλληλα, άρθρο 160, παραπομπή παράλληλα στο άρθρο 160, κεφάλαιο 10 της συνθήκης, το οποίο αφορά την κοινωνική πολιτική. Τώρα, όσο αφορά τα στοιχεία ε, στα οποία θα ήθελα να επανέλθω. Ζητώ συγγνώμη, γιατί έχω συντάξει ήδη έναν κατάλογο και θα τον συμβουλευτώ, αλλά αυτό θα με βοηθήσει να είμαι πιο συγκεκριμένη. Πρώτον, κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας υπήρχε μία ε, επιθυμία ε, των δικτών, ε, επεξεργασίας μιας εργαλειοθήκης που θα εξόπλιζε την, ε, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στις συζητήσεις με την ΕΚΟΦΗΝ. Θεωρείτε ότι αυτό η, η δουλειά εγκαταλείφθηκε ή αντίθετα ε, βασίζεστε ή, ή επί τη βάση αυτής της εργασίας είναι που η Επιτροπή μπόρεσε να προχωρήσει στην εξειδίκευση κάποιων δικτών. Θεωρείτε ότι αυτή είναι η καλή στρατηγική. Ε, συνεχίζω στο θέμα των δικτών. θεωρείτε ότι πέρα από την δουλειά που κάνετε εσείς, εάν θέλουμε οι δείκτες αυτοί να είναι ε, κατάλληλοι, σωστοί, να, να περιέχουν πραγματικά τα στοιχεία της προηγούμενης περίοδου, ε, δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο να κληθούν και οι κοινωνικοί εταίροι ε, να συμμετέχουν στην εκπόνηση αυτών των δικτών. Μιας και μιλάμε για κοινωνικό διάλογο, νομίζω ότι αυτή η στρατηγική ε, είναι κερδοφόρα για όλους. Ο κύριος ε, Τομάς Ντομινίκ μίλησε για τους δείκτες. Εμάς μας ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που είπε ο Επίτροπος στον τομέα αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ. Υπάρχει μια πραγματική εξέλιξη. Ε, υπάρχουν περιθώρια να πιστεί το Συμβούλιο καθώς και το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Τρίτον, ε, μία ερώτηση προς τον κύριο Τόμ Μπέβερς κατά την ετήσια εξέταση της, ε, της ανάπτυξης, ίσως να μην γνωρίζετε ότι υπάρχει μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας καλώ να την εξετάσετε προσεκτικά. Να δείτε με την προσέγγιση που εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε εδώ ε, το, στο Κοινοβούλιο θα δείτε ότι έχουμε μια γενική οπτική η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην οπτική της Κομισιόν και προσπαθούμε να επιφέρουμε μια προστιθέμενη αξία, μια πρόσθετη αξία. Ε, και αν δεν το κάνω εγώ, δεν επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή τη γνωμοδότηση, κανείς δεν θα το κάνει άλλος. Τέταρτον αναθεωρήσατε το 1 τρίτο των συστάσεων αναχώρα. Αυτό ε, προήλθε από την πλευρά του κεφαλαίου, προήλθε από την, μια, ένα αίτημα της ε, Κομισιόν να αναθεωρηθούν ε, οι, να αναθεωρηθεί ο κοινωνικός πυλώνας. Δεν θα έπρεπε να έρθουν και εδώ οι κοινωνικοί εταίροι. Ε, από τότε που προεδρεύω αυτή της Επιτροπής παρατηρώ μια απουσία κοινωνικού διαλόγου. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή και η... Η ΕΚΟΣΟΚ έχει ζητήσει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. και σας θυμίζω και την ιστορική μας κληρονομιά, τον Ζακ Ντελόγ, τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια διάσταση που πραγματικά λείπει. Ε, Ούτε και η Τρόικα δεν το έχει κάνει. Αυτό το λογικό στοιχείο του, του, του κοινωνικού διαλόγου λείπει. Έκτον, Όσο αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, επιτρέψτε μου λίγο να εξηγήσω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί μιας και τώρα εφαρμόζουμε τις πολιτικές αυτές, να περάσει αυτό το μήνυμα. Υπάρχει μια βούληση το ΕΜΚΟ ε, να μπορέσει να περάσει το μήνυμα και να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις στον συντονισμό. Εμείς πάλι θέλουμε να υπάρχει ένας χώρος δημιουργικότητας, να υπάρχει να μπορέσουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να ανταλλάξουν τις καλές τους πρακτικές, ε, να, να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά να πάρουμε εκείνες τις μορφές κοινωνικής προστασίας που υπάρχουν και λειτουργούν και να τις επεκτείνουμε. Εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια δίωδος ε, για να περνούν οι προτάσεις από τη μία στην άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ποιο, ποιος είναι ο απολογισμός. Εν τέλει, είπατε ε, μιλήσατε για τις κατευθυντήριες γραμμές για την εργασία που πρέπει να αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Ε, εγώ φυσικά είμαι υπέρ ε, των γενικών κατευθύνσεων από, χρόνων. Είμαι υπέρ. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές μαζί να τις αναπτύσσουμε ούτε ότι όλες είναι της ίδιας σημασίας. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα προνομιούχα εργαλεία, τα προνομιακά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη, τι μπορεί να μας φέρει. Ε, νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο, η σημασία της έχει χαθεί, μάλλον η σημασία των κατευθυντήριων γραμμών έχει χαθεί λίγο. Αν μήπως είναι δύο εργαλεία που έχουν τελικά τον ίδιο σκοπό. Από την αρχή, δηλαδή από το 2009-10, η Κομισιόν δεν θεώρησε ποτέ ότι οι κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης θα όφυλαν να μεταβάλλονται. Ενώ στον ενώ πραγματικά συμβαίνουν κοσμοϊστορικά πράγματα στον τομέα της ε, απασχόλησης. De, de, euh, de ε, ε, εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτά τα εργαλεία. Τι θα κάνουμε με αυτά τα εργαλεία. Είναι αμετακίνητα από τη στιγμή που τα υιοθετήσαμε ή πρόκειται να τα προσαρμόσουμε και να τα αξιοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το διάλογο μεταξύ των θεσμών και των οργάνων. Ε, είναι 12.30, ο διάλογος έχει τελειώσει. Ε, ευχαριστώ τους ε, διερμηνές, τους διερμηνείς για την υπομονή τους. Δεν είναι καλή αρχή για το 2014. Ο καθένας έχει πέντε λεπτά με διερμηνία για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλια και τις προτάσεις. Είναι πολύ δύσκολο μέσα ένα πεντάλεπτο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα δώσω κάποιες γενικές απαντήσεις. Καταρχήν, τι μαθήματα διδαχθήκαμε από την κρίση και τι μαθήματα διδαχθήκαμε από τις κοινωνικές πολιτικές. Η, η Επιτροπή μας αναλύει τις εξελίξεις των μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη και συντάξαμε και έναν πίνακα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Θα ήθελα απλώς να διαβάσω τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Τα αποτελέσματα λοιπόν, τα συμπεράσματα λένε τα εξή. Τα κράτη που εφαρμόζουν προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίασης ε, έδειξαν μεγάλη προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να, να αντλήσουμε κάποια μαθήματα από τις εμπειρίες. Θα πρέπει να ε, ε, ε, ενισχυθούν τα, προβλήματα, τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν έγινε προσπάθεια πολέμηση της φτώχειας. Ε, ε, θα πρέπει μερικές επιπτώσεις να μελετηθούν πριν την εφαρμογή των δημοσιονομικών προγραμμάτων ανάλογα με τι ομάδε ηλικιακέ και τι ομάδε οδήματο. Οπότε τα συμβούλια, το Συμβούλιο τακτικά θα πρέπει να κάνει ε, μια αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών Κοινωνική Πολιτική με τα προγράμματα οικονομική προσαρμογή, προκειμένου να δώσει κάποιε ε, προσανατολισμούς πολιτικής. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα τη έκθεσή μα και αυτό ήταν ένα από τα μαθήματα που αντλήσαμε ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε μεταρρύθμισης και οποιοδήποτε προγράμματος προσαρμογής οικονομικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις. Να δώσω και εγώ κάποιες απαντήσεις εκ μέρους της δικής μου επιτροπής. Καταρχήν ως προς τα λάθη που έκαναν τα κράτη-μέλη. Ε, και τα λάθη στις, ε, οικονομικές, στις κοινωνικές πολιτικές και τις κοινωνικές απασχόλησεις. Εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη κάνουν λάθος, απλώς ε, οι πολιτικές επιδέχονται βελτιώσεις και οι ειδικές συστάσεις αναχώρα δίνουν κάποιες προσανατολισμούς και κατευθυντήριες γραμμές. Είναι σημαντικά τα μεταρρυθμιστικά πακέτα και είναι εύκολο να λαμβάνει κανείς το λόγο μετά το ρεμοντόρες, γιατί κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, οικονομικές και δημοσιονομικές θα πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις της ε, αγοράς εργασίας προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοχή των μεταρρυθμίσεων από τους κοινωνικούς εταίρους και να βελτιώνεται και η αποτελεσματικότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και φυσικά να υιοθετηθεί μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που θα γίνει αντιληπτή από την κοινωνία, όπως είπε και ο κύριος Τόρες. Σας ευχαριστώ που υπενθυμίσατε το ρόλο που μας κατοχυρώνει η συνθήκη και ο ρόλος μας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών αλλά και η συνεργασία με την Επιτροπή ΕΚΟΦΗΝ για την ε, οικονομική πολιτική. Έχουμε αγαστή συνεργασία και με την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚΟΦΗΝ και προσπαθούμε όταν συντάσσουμε τα, τις ειδικέ στάσεις από την αναχώρα να εξετάζουμε τα διάφορα προβλήματα και να λαμβάνουμε υπόψη τις κοινέ ανησυχίε. και προσπαθούμε να έχουμε μια συντονισμένη θέση του Συμβουλίου σε επίπεδο Επιτροπής ώστε όλες, ε, όλοι οι φορείς πολιτικής να βρίσκονται προς την ίδια κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες, σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια για το έργο της Βελγικής Προεδρίας γιατί ως Βέλγος ε, και ως πρόεδρος ε, το, της ε, ομάδας εργασίας για τους δείκτες. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Επίσης είχα, έχουμε και τον δείκτη επιδόσεων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής απόδοσης. Είναι πολύ σημαντική αυτή οι δίκτες γιατί οι αγορές εργασίας είναι περίπλοκα συστήματα και δεν μπορούμε να συνοψίσουμε την κατάσταση με λίγους δείκτες. Πάντως ο δίκτυς ε, επιδόσεων είναι πολύ σημαντικός ε, για επικοινωνιακούς λόγους. Μπορεί να μην είναι ιδεώδης. Ο πίνακας των επιδόσεων, το scoreboard, ε, είναι συμπληρωματικός. Τον συνδυάζουμε με το δίκτυο επιδόσεων κοινωνικής προστασίας, ώστε να έχουμε ένα συνεκτικό πλέγμα δικτών. Σε ό,τι αφορά το μέλλον του πίνακα του scoreboard, θα το συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους που ήδη έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και συμφωνούμε με τους κοινωνικούς εταίρους ε, ότι είναι σημαντικό να γίνουν διαβουλεύσεις μαζί τους. Σας ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις σας, ότι θα πρέπει στο μέλλον ε, να, έχουμε πιο στενές διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη έχουμε νομίζω κοινό ενδιαφέρον για μια σφαιρική προσέγγιση, μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι ειδική θεώρηση ανακράτος μέλος. Συμφωνούμε με αυτή τη σφαιρική προσέγγιση. Επίσης ρωτήσατε τι γίνεται με τις ειδικές ανά αναχώρα και με τις τροποποιήσεις που κάνουμε. Το σημείο αφετηρίας ε, είναι ότι ε, το κράτος μέλος που λαμβάνει τις στάσεις θέλει κάτι να αλλάξει. Αλλά εμείς ως Επιτροπή φροντίζουμε να τις εξετάζουμε με πολυμερή τρόπο. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε τις ε, γνωμοδοτήσεις και την εμπειρία των 27 άλλων χωρών, άλλων χωρών, συγγνώμη, όλες οι χώρες εξετάζουν ε, τις συστάσεις. Δεν είναι διμερής ε, συζήτηση μεταξύ του κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης έχουμε πολυμερή εποπτεία και τα συμπεράσματα της πολυμερούς εποπτείας είναι το σημείο αφετηρίας για την γνωμοδότηση της ΕΜΚΟ, της δικής μας Επιτροπής για τις ε, συστάσεις αναχώρα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε πολλές περιπτώσεις εμείς ε, ε, ακολουθήσαμε διαφορετική άγουσα, είτε διαφορετική από την Επιτροπή, είτε διαφορετική από το κράτος μέλος. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως η δημιουργικότητα, η ευρηματικότητα θα πρέπει να είναι η βάση και να επιτρέψουμε ανταλλαγή πρακτικών στο δίκτυο. Εκεί η ΕΜΚΟ θα έχει ρόλο παρατηρητή. Δεν θα πρέπει να προσδιορίσουμε δηλαδή ένα σημείο αφετηρίας προσδιορίζοντας από την αρχή το έργο του δικτύου. Πάντως η εμπειρία μας, κυρίως από τον κοινωνικό διάλογο, μας έχει διδάξει ότι αν δεν δημιουργήσουμε δεσμούς μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και των διαφόρων σταδίων της ίδιας διαδικασίας, θα περιπλέξουμε υπερβολικά τα πράγματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη ροή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Γι' αυτό θέλουμε το ρόλο παρατηρητή στο δίκτυο. Και τέλος για τους κοινωνικούς εταίρους ναι, πολλές συζητήσεις έγιναν και εμείς ε, συμφωνούμε με τις ενώσεις κοινωνικών εταίρων και τις οργανώσεις τους ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και μάλιστα ε, η βελτίωση αυτή θα πρέπει να φανεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η συμμετοχή του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, για τις κατευθυντήρες γραμμές, είπατε ότι είναι κοινό συμφέρον και της Επιτροπής μου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τις αναζωογονήσουμε γιατί καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερο λόγο για τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση από ό,τι έχουμε για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη που είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε νέα πνοή και σε αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στη συνθήκη θα έπρεπε να είναι ισχυρότερο από αυτό το, το οποίο ε, αποτελεί την πρακτική. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει η Πρόεδρος, τους διερμηνείς, διότι μας συνόδευσαν μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης και εμείς ευχαριστούμε τη σειρά μας. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή τους, λέει η Πρόεδρος. Και θα ήθελα μετά από την πρωινή μας συνεδρίαση να ζητήσω και να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά, να επαναληφθεί και να αποκατασταθεί αυτή η πρακτική ε, της ε, ακρόασης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι κάτι που βοηθάει όλους μας. Σας ευχαριστώ όλους έχει ολοκληρώσει η εξέταση της ημερήσιας διάταξης. Επόμενη συνεδρίαση στις 22 Ιανουαρίου. Συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια το πρωί της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ όλους και όλες. Θα τα πούμε εκεί.